Mes chers collègues, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σα. Commençons. Πάμε. Πάμε. Ισμαήλ Ερτούγκ. Είπα ότι αρχίζει η συνεδρίαση. Αλλά πριν αρχίσουμε, θέλω να χαιρετήσω τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας. Ευτυχώς που σας έχουμε για να εξασφαλίζεται και η Ένωση στην πολυμορφία. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε το μήνυμα των διερμηνέων. Οι διερμηνείς έχουν το λόγο. Βρισκόμαστε στην 35η μέρα των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των συνθηκών εργασίας που επέβαλε η μερα των κινητοποιησεων διαμαρτυρια κατα των συνθηκων εργασια που επεβαλε η διοικηση στου διερμηνεί. Συνεπώ δεν θα παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου για την παρούσα συνεδρίαση που θα τελειώσει ακριβώ την προγραμματισμένη ώρα η διερμηνία. Σα ευχαριστούμε για την προσοχή σα.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 Merci Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα αυτό. Δεν σας ακούω τη γαλλική διερμηνία τώρα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, τώρα εντάξει, πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Πάμε λοιπόν. Έγκριση μερίσια διάταξη, Αν δεν έχετε αντιρρήσει. μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένο το σχέδιο μερίσια διάταξη, Πολύ ωραία πρακτικά των συνεδριάσεων της 7ης Ιουνίου καθώς επίσης και της 20ης και 21ης Ιουνίου μπορούν να εγκριθούν αν δεν έχετε αντιρρήσει και πάλι που δεν έχετε από ό,τι βλέπω. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Γνωρίζετε όπως και εγώ ότι η Ολομέλεια απέριψε τις τρεις κοινωνικές ε, προτάσεις της δέσμευσης μέτρων για την κινητικότητα προς ενημέρωση σας ανακοινώνω ότι θα το συζητήσουν οι συντονιστές αργότερα σήμερα. Περνούμε λοιπόν αμέσως στο πρώτο θέμα μας, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Όλα τα τμήματα. Ο κύριος Τέλιτσκα είναι ο συγκητής μας. Και μετά θα προσπαθήσω να αρχίσει και η συζήτηση. Καλή σας μέρα κύριε Τελίτσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιες ιδέες εδώ. Ο προπολογισμό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά σταθερός. Βεβαίως δυσκολίες θα προκύψουν όταν θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να θυμίσω στην Επιτροπή Τραν τι σημαίνει σταθερότητα στον προπολογισμό και τι είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να περιμένουμε. Τα βασικά σημεία που θέλουμε να διαφυλάξουμε είναι οι περικοπές στο ΕΦΣΥ, τα προγράμματα χρηματοδότησης που θα εκπνεύσουν. Οι επενδυτές χρειάζονται σταθερότητα για τη χρηματοδότησή του εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια, ο οργανισμός η, όπως η ΆΣΑ, η ΕΝΙΣΑ έχουν δει την εντολή τους να παρατείνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζονται και αρκετού πόρους για να υπάρξει συνέχεια στο έργο τους. Για μεγάλο μέρο ούτω ή άλλω τη υλοποίηση ε, του κεκτημένου, νομικού κεκτημένου, χρειάζεται η συνεργασία του. Ε, για ε, τι κοινέ επιχειρήσει όπω το ΣΕΖΑΡ, χρειάζεται πάλι και η δική του συνέχεια. Δεν θα Η δική του συνδρομή δεν θα μπορέσουμε εδώ να συμβιβαστούμε. Και θα περιμένουμε και την ε, ε, θέση σε λειτουργία 8 δορυφόρων εδώ για τον ίδιο σκοπό. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε στα βασικά και δύο σημεία στα οποία σίγουρα δεν θα διαφωνήσουμε. σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό μεταφορών, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το 2019 είναι το τελευταίο δημοσιονομικό έτος της θητείας. Και θα υπάρξει υλοποίηση των περισσότερων προγραμμάτων μέχρι τις εκλογές για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπροασκευαστικές δράσεις. Για τελευταία φορά στη θητεία μας έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε οικονομική συνδρομή σε προγράμματα που πρέπει να συνδεθούν απευθείας με τις πολιτικές μας προτεραιότητες και τα νομοθετικά ντοσχεία που αυτή τη στιγμή μελετούμε. Αυτά είναι τα κριτήρια και οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή των προγραμμάτων που θα υποβάλουμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για να αποφασίσει. Από δική μας πλευράς θα σας παρακαλέσω να με βοηθήσετε ώστε να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Και το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω και λογικά συνδέεται με τα προηγούμενα είναι η δημοσιονομική γραμμή που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Σε σχέση με άλλα θα μπορούσε καλής να πει ότι είναι αρκετά περιορισμένο, αλλά Έχουμε δυσκολία στις ευρωπαϊκές μεταφορές σε ένα κόσμο ψευδών ειδήσεων. Ο κόσμος δεν ξέρει αρκετά για τα δικαιώματά του. Εάν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, ο κόσμος μπορεί να ε, λάβει γνώση των δικαιωμάτων του και να μπορεί μετά και να τα ασκήσει. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε, να ασχοληθούμε με την έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υπάρχει για το θέμα αυτό. Τα δικαιώματα των επιβατών είναι κάτι που πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα και να είναι περιτά. Είναι ξεκάθαρη εικόνα, τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Έχουμε και εισηγητή από την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι οι ανάγκες των μεταφορών θα αντικατοπτριστούν επαρκώς στις διαπραγματεύσεις. Και βάσει αυτών των γραμμών σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Τέλιτσκα. Ξεκινάει η συζήτηση. Κύριε Σαλίνη. Ευχαριστώ. Ε, οι γνώμη μας ως ομάδας και η δική μου προσωπικά είναι ότι οι γραμμές του εισηγητή είναι απολύτως συνεπείς. Και με τη δική μας άποψη για το τι προτεραιότητες θα πρέπει να έχει ο προπολογισμό ε, για τις μεταφορές και για τον εντοπισμό της σημασίας του τομέα των μεταφορών ως προς την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη οι απόψεις που αναπτύσσει ο εισηγητής γύρω από τα θέματα αυτά είναι απόψεις με τις οποίες συμφωνούμε απολύτως. Ε, για συγκεκριμένες παρατηρήσεις, πριν φτάσω στα πιλωτικά προγράμματα, οι μεγάλες ε, προτεραιότητες για μας είναι το ΣΕΦ πρώτα απ' όλα, η διευκόλυνση διασύνδεσης της Ευρώπης. Εδώ πρέπει να πηγαίνουν αρκετά κονδύλια στο πρόγραμμα αυτό, του οποίου τα αποτελέσματα τα επιβεβαιώνει και η εκθεσή μας. Ε, εδώ δεν έχουμε καμία επιλογή. Δεν μπορούμε να περικόψουμε τα κονδύλια του προγράμματος αυτού. Το αντίθετο και για άλλους οργανισμούς, για την ΕΑΖΑ και την ε, ΕΝΙΣΑ, συμφωνούμε το Τα κονδύλια που προορίζονται για τους οργανισμούς αυτούς πρέπει να αναλογούν και στην σημασία τους, δηλαδή να ενισχυθούν. Στο σημείο 3, πολύ γρήγορα, Η στρατηγική σημασία των Γαλιλαίο και Έγνος για την διαστημική μας πολιτική είναι σημαντικά και για τον οργανισμό του διαστήματος. Συμφωνώ εδώ λοιπόν με τον εισηγητή Τελίτσκα και μετά και στο τέταρτο για τα μακρολήματα, για να το πω έτσι, του προπολογισμού, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το Sky και το ΣΕΖΑΡ είναι επίση προγράμματα που πρέπει να υποστηριχθούν. Στο τέταρτο τώρα κεφάλαιο τη έκθεση ε, για τα πιλωτικά προγράμματα, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι έχουμε ε, μελετήσει με προσοχή όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι ε, σκοπεύει να επιδιώξει, αλλά θα πρέπει για συγκεκριμένα στοιχεία του, των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων να διατηρήσουμε ένα περιθώριο διότι έχει κάνει κάποιους υπολογισμούς η Επιτροπή και γενικώ συμφωνούμε. Υπάρχουν όμως και προγράμματα που θα πρέπει να τα δούμε επιμέρους για να υπάρχει και συμφωνία ε, με το γενικό πνεύμα που θέλουμε να διέπει τον προπολογισμό και να δούμε ποιε είναι και οι συγκεκριμένε προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Πάντω, γενικώ η δουλειά που έχει γίνει είναι εξαιρετική, θεωρώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, ε, Ο κύριο Βαντάλεν. αντικαθιστάτε τον κύριο Ζήλε, όχι. Η κυρία Ντερμόντε αποσιάζει, άρα θα την εκπροσωπήσει ο κύριο Σερτόκ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου ε, τη συναδέλφου Ντεμόντε γιατί βρίσκεται καθόλου προ τι ε, Βρυξέλλε. Νομίζω πω πετάει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να παρουσιάσω τη δική τη τοποθέτηση σε σχέση με αυτήν την ε, πρόταση ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Τέλτσκα για αυτή την αξιέπαινη δουλειά που έχει κάνει σε σχέση με αυτό το περίπλοκο φάκελο. Γιατί βέβαια η σχετική πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για την συνολική ανταγωνιστικότητα αλλά και την εδαφική συνοχή τη Ευρώπη. Άρα λοιπόν η πολιτική μεταφορά χρήζει και ενό φιλόδοξου προπολογισμού, ο οποίο θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε ε, των προγραμμάτων και των ε, project που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βέβαια μιλάμε για έργα υποδομή, χρειαζόμαστε ε, υψηλά, υψηλού, υψηλά ποσά και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου. Και γι' αυτό λοιπόν είναι εξαιρετική σημασία να σταματήσουν οι περικοπέ ε, του προπολογισμού για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΣΕΒ, ε, όπω έγινε κατά τελευταία χρόνια, προκειμένου να έχουμε περαιτέρω κίνητα για το πρόγραμμα. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν την δέσμευση τη Επιτροπή για αύξηση κατά 39,4 και 5,3 αντιστοίχω των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, αλλά η εν λόγω αύξηση δεν είναι επαρκή αν λάβουμε υπόψη μα τι περικοπέ που έγιναν στο παρελθόν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτό αυτά τα κονδύλια αξιοποιούνται με τον τρόπο εκείνο που θα επιτρέψει τουλάχιστον ε, ε, την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του δικτύου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτύχουμε την σωστή εφαρμογή των σχετικών έργων. Δυστυχώ δεν υπάρχει το απαρκέ ενδιαφέρον από πλευρά τη Επιτροπή ε, για τον Τουρισμό, παρότι αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο οικονομικό κλάδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λάβει ε, περισσότερη σημασία και μια ξεχωριστή γραμμή του υπροπολογισμού που θα οδηγήσει σε περισσότερη διαφάνεια αλλά και ανάληψη των εθνών από την πλευρά τη επιτροπη σε ό,τι αφορά τι επενδυσει σε αυτό το τομέα, τον τουρισμό. Πολύ. Ο ε, επόμενο ε, Thank ευχαριστώ. Η πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετική σημασία για την οικονομική, ε, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα προκειμένου να διευρυνθεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιώσιμο τρόπο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της συγχρηματοδότησης σε ό,τι αφορά ε, την βελτίωση του συνδρομικού δικτύου και εδώ θα πρέπει, ε, θα πρέπει να ε, τονίσουμε την μετάβαση που θα γίνει προς πιο βιώσιμού τρόπου μεταφορών. Ευχαριστώ. Κυρία Κίλονεν, εσείς αντικαθιστάτε την κυρία Λόπες, όχι. Ε, τότε η κυρία Άντερσον, Θα ήθελα απλώς να χαιρετήσω τη δουλειά που έχει γίνει σε σχέση ε, με αυτό το βάτελο και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Τελίσκα σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα των επιβατών και το γεγονό ότι δεν υπάρχει επαρκή ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα δικαιώματα. Και πέρυσι ε, το ελεγκτικό συνέδριο πράγματι διαπίστωσε ότι υπάρχει εδώ μεγάλη στέρηση σε ό,τι αφορά δηλαδή την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ω επιβάτε. Θα πρέπει να γίνει κάτι εδώ γιατί μόνο το 1 τρίτο των Ευρωπαίων τελικά γνωρίζει το πλαίσιο σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και θα πρέπει να σημειωθεί αυτό. Και νομίζω πω σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να κάνουμε λόγο και για ένα πανευρωπαϊκό έντυπο για την υποβολή παραπώνων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει και έχει λάβει και την υποστήριξη από πολλέ πλευρέ. Ευχαριστώ. Θα σα ξαναδώσω το λόγο κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Να τονίσω μόνο τα εξή δύο σημεία που προέκυψαν και από τη συζήτηση. Ο κύριος Σαλίνη μίλησε για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι ε, η γενικότερη στόχη. Επίσης μου άρεσε και αυτό που άκουσα πάλι από τον κύριο Σαλίνη για την αξιολόγηση των πιλωτικών προγραμμάτων. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει βέβαια να ακούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει εμπειρογνωμοσύνη και κάνει κάποια αξιολόγηση, αλλά και εμείς έχουμε ίδια γνώμη. Και στο παρελθόν ε, κάποιος είχε προωθήσει ένα σχέδιο, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ποιος ήταν αυτός, ε, και ε, το εγκρίναμε και την επόμενη μέρα εμφανίστηκε ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κεντρική ιδέα και η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι υποστηρίζουμε ε, τις ε, προτεραιότητες πολιτικής που έχουμε ιδιαίτερα στο τελευταίο οικονομικό έτος ε, της δικής μας θητείας. Συμφωνούμε περισσότερο αυτή τη φορά, έχουμε περισσότερη συνοχή από ανταγωνισμό μεταξύ μας και χαίρομαι γι' αυτό και το εκτιμώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τελίτσκα. Σας έδωσα το λόγο διότι ήθελα να ξανακούσω ε, την άποψή σας και ξέχασα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη σημασία σας δίνω. Η κυρία Αν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Σιγητά, θα προσπαθήσω μόνο να προσθέσω μερικά σημεία στα θέματα και τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Ε, είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός μεν, όπως ε, ακούσαμε. Και ε, βασίζεται σε μια ανάλυση που κάνει ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον οργανισμό που λαμβάνει υπόψη ε, όλα τα συμβόλαια και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Δηλαδή οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα ε, συνδέεται με προβλήματα για την εκταμείωση των κοδηλίων προς τους δικαίουχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καλωσορίζει και χαιρετίζει το ψήφισμα για τον προπολογισμό σας. Επίσης, τονίζεται και την ε, προκήρυξη που έχει γίνει φέτος ε, για να δαπανηθούν τα κονδύλια της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη, και να καλύψουμε το κενό και την καθυστέρηση του παρελθόντος. Τώρα, για τα παλιά προγράμματα επίσης θα προκηρυχθεί ε, η ανάκτηση των κονδυλίων από προγράμματα του παρελθόντος, 80 εκατομμύρια τα υπολογίζουμε σήμερα, να δούμε του χρόνου αν θα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καιρό συζητεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε μήπως μπορούμε να προκηρύξουμε ε, μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το μέσο ΣΕΦ. Όταν θα έχουμε ε, νέες προτάσεις μπορεί να έρθουμε να σας τις παρουσιάσουμε το φθινόπωρο. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό των ευρωπαϊκών οργανισμών. Ξέρω πόσο υποστηρίζει το κοινοβούλιο σας τον προπολογισμό. Για τον ε, Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Οργανισμό δεν μειώνεται ε, ο προπολογισμό, διότι το 2019 κανονικά είναι το έτος κατά τον οποίο τα τέλη θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και έχει εγγράψει στον προπολογισμό του οργανισμού 3,8 εκατομμύρια ευρώ που θα προκύψουν από τα τέλη που θα εισπράξει. Άρα είναι λίγο μικρότερη η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, αυξάνεται η συνολική τους χρηματοδότηση ε, χάρη ε, στα τέλη που θα αρχίσουν να εισπράττουν από το 19. Και για τα πιλωτικά προγράμματα σημείωσα τις παρατηρήσεις σας. Στο παρόν στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες πρώτες αξιολογήσεις. Βεβαίως, τις οριστικές θα τις λάβετε εν ευθέτω χρόνο, όταν θα ε, δημοσιευθεί η επιστολή ε, εκτελεσιμότητας. Πάντως, το Σεπτέμβριο. Ε, τα περισσότερα τα υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μοντανιό. Θυμίζω την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 13 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Οι ε, βουλευτές μπορούν να κάνουν δύο τροπολογίες, μία τροπολογία στο σχέδιο, δύο ειδών τροπολογίες μάλλον, δημοσιονομικές και για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και κανονικές τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης. Περνούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Χουντάκ, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με θέμα τη χρηματοδότηση των μεταφορών. Θα τον υποδεχτούμε. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή μου. Allez-y, prenez place. Alors, monsieur Dac, nous avons... Κύριε Ουρντάκ, σας έχουμε προσκαλέσει για μια ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ σε σχέση με τον κλάδο των μεταφορών και σας καλωσορίζω. Είναι επίκαιρη και σκόπιμη η συζήτησή μας σήμερα διότι από τη μία υπάρχουν οι ανάγκες για επενδύσεις για να εξυγχρονιστούν οι μεταφορές μας, αλλά και να διαμορφώσουμε τις μεταφορές για το μέλλον σε σχέση και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, την ψηφιακή επανάσταση, ψηφιοποίηση και στις μεταφορές, κλιματικές αλλαγές. Εδώ θα χρειαστεί πραγματικά ενεργειακή μετάβαση. Από τη μια λοιπόν επιτάπητος έχουμε τα επόμενα προγράμματα όπως τον, ε, τη διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης και ε, τα επόμενα προγράμματα στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και περιμένουμε να μας πείτε σήμερα ποιες είναι οι δικές σας απόψεις για τα θέματα αυτά. Ποιες είναι οι προοπτικές και τι είδου έργα θα επιλέξετε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα ή τέλο πάντων να τις επιδιώξουμε. Θα σας δώσω το λόγο για κανένα δεκάλεπτο και μετά θα έχουμε συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να σας μιλήσω για τη δουλειά της ΕΤΕΠ στον τομέα των μεταφορών. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Θυμάμαι λίγο τη δουλειά μου στην κυβέρνησή μου όταν ήμουν Υπουργό Οικονομικών και έπρεπε να πηγαίνω στο, στις Εθνικές Βουλές και με, ψή, με και έπρεπε να περάσω τα πάνδυνα για να απαντήσω στον ε, τομέα των ε, μεταφορών τώρα. Πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά την ΕΤΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, ανήκουμε στα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακολουθούμε και τι στρατηγικέ και τι πολιτικέ του προτεραιότητε. Αυτέ τη Ένωση δηλαδή. Ενημερωτικά, φέτο γιορτάζουμε τα 60 χρόνια ε, λειτουργία τη ΕΤΕΠ, ένα μέρο ε, ευρωπαϊκή ιστορία για το οποίο μπορούμε να είμαστε και υπερήφανοι, διότι η ΕΤΕΠ από το 1958 εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παγκοσμίω. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι για κάποια πράγματα. Συγκριτικά, πέρσι χρηματοδοτήσαμε έργα και προγράμματα με 80 δις ευρώ. Η Παγκόσμια Τράπεζα σε τη διαστολή έφτασε τα 60 δις επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι για την Ευρώπη κάνουμε πολλά καλά. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τομέα των μεταφορών, είναι από τις προτεραιότητές μας. Κατά μέσο όρο, ετησίως ε, αποδίδουμε 13 δις σε έργα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλαμβάνονται και κάποια έργα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δέκατο των δραστηριοτήτων μας είναι εκτός Ένωσης, ιδίω στις χώρες της γειτονία. Το πρωί, για παράδειγμα, υπέγραψα σύμβαση έργου με αναπληρωτή υπουργό, υφυπουργό τη Ουκρανία για την ε, οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των οδικών μεταφορών στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό τα έργα μα να διαδίδουν και τι ευρωπαϊκέ αξίε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στι χώρε τη γειτονία. Τα 13 δις λοιπόν είναι το κατά προσέγγιση μέγεθος των επενδύσεών μας, 17% του συνόλου των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ. τριών λογιών δραστηριότητες έχουμε, το lending, το blending και τη συμβουλευτική. Η δανειοδότηση θα πει ότι έχουμε συνεννοήσεις με κυβερνήσεις, με ιδιωτικό τομέα, με πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Η, το blending, η ανάμειξη, είναι αυτό που αναφέρετε και εσείς πρόεδρε, όταν λέγαμε για τη διευκόλυνση διασύνδεσης της Ευρώπης δηλαδή ε, με συνδυασμό δωρεών, ε, κλασικών διαρθρωτικών ε, κονδυλίων, ποσά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Κοιτάζουμε ποια ποσά μπορούμε να συνδυάσουμε και τι μπορεί να επιστραφεί και να υποστηριχθεί και από ιδιωτικά ποσά. Και η συμβουλευτική θα πει ότι έχουμε σημαντικό όγκο επιχειρήσεων. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με κυβερνήσει, με εθνικού και τοπικού φορεί, με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να έχουμε την κατάλληλη παρακολούθηση των προγραμμάτων μα αυτού του είδους τις δραστηριότητε αναπτύσσουμε. Εάν δούμε τις υποδομές των μεταφορών συνολικά στην Ευρώπη, εμείς βλέπουμε ότι ιστορικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1% του ΑΕΠ πήγαινε στις μεταφορές ούτως ή άλλως. Ο αριθμός αυτός έτεινε να φύνει σε περίοδο, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και τώρα βλέπουμε στις μεταφορές στην Ευρώπη να υπάρχει ένα μια τάση να αυξηθούν. Αν δείτε τους αριθμούς, οι συντονιστές για τις μεταφορές υπολέξαν ότι για το επόμενο πουδουπού αυτό το χάσμα στις επενδύσεις θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο, μόνο και μόνο για τους διαδρόμους TNT. Εάν δείτε το συνολικό μέγεθος, μιλάμε για 200 δις ευρώ και όχι εκατομμύρια. Ε, χάσμα 200 δις ευρώ που θα πρέπει να καλυφθεί ε, ως προς τις επενδύσεις μας στις υποδομές των μεταφορών. Έχουμε λοιπόν σημαντικό ρόλο εδώ να διαδραματίσουμε και πολλά πρέπει να γίνουν. Εξετάζουμε όχι μόνο τις παραδοσιακές υποδομέ των μεταφορών, ιδίω τους διαδρόμου TNT, γιατί είμαστε ευρωπαϊκές τράπεζες και κοιτάζουμε τα έργα στις μεταφορές που έχουν ε, ένα, μια δυνατότητα να παράγοντα διασύνδεσης, αλλά και νέους τρόπους μεταφοράς. Ε, βιώσιμες μεταφορές, καθαρότερες και με χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει τη διευκόλυνση ε, καθαρότερων μεταφορών για να ενισχύσει τα σχετικά τεχνολογικά μέσα σε πόλεις όπως η Καρτουά, η Λασπάλμας. Ε, χρηματοδοτήσαμε εκεί δίκτυα λεωφορείων που χρησιμοποιούν ε, καθαρή ενέργεια ή και νέες υποδομές στα πλαίσια ε, ηλεκτρονικής ε, μορφής, στα πλαίσια των διαδρόμων TNT. Αυτά για να συνδυάσουμε στόχους της ψηφιοποίησης, του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Όπως ξέρετε η ΕΤΕΠ ασχολείται με την εκτέλεση του ΕΦΣΥ και μπορώ να σας πω ότι ως το τέλος Ιουλίου το ποσό για την πρώτη περίοδο του ΕΦΣΙ 315 δις με τις εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και της ε, ΕΤΕΠ θα έχει πετύχει πολλά. Για μας είναι ξεκάθαρη η επιτυχία το ΕΦΣΙ και αποδεικνύει ότι τα κενά στις επενδύσεις δεν μπορούν να καλύπτονται μόνο από κρατικά κονδύλια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε ενίσχυση, μόχλευση και από ιδιωτικού πόρου. Το ΕΦΣ είναι ένα τρόπο να γίνει. Γι' αυτό η όλη προσπάθεια είναι πολύ σημαντική και για την ΕΤΕΠ. Στο μέλλον και βλέποντας και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τη συνιστόσα InvestEU, βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί το ΕΦΣΙ και ήδη συζητάμε τις ε, ερωτήσεις μας για το πώς ακριβώς θα διαρθρωθεί το InvestEU. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια τη συζήτησή μα. Τώρα για το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Ε, Ω τώρα έχουμε υποστηρίξει 59 έργα για τι μεταφορέ που υποστηρίζει η εγγύηση του ΕΦΣΙ και θα κινητοποιήσουν 25 δις ε, παρελκόμενων επενδύσεων. 8% του συνολικού όγκου του ΕΦΣΙ γέννηση της επενδύσεις μεταφορών λοιπόν. Γιατί μόνο 8%? Γιατί χρειάζεται και ένα στοιχείο ιδιωτικού τομέα στο ΕΦΣΥ. Και ε, οι υποδομέ των μεταφορών στην Ευρώπη χρειάζονται και ένα σκέλο ε, συμβάσεων, εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Για να λειτουργήσουν και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο έργων έχουμε ασχοληθεί και με την εταιρεία μεταφορών της Ρήγα στην Λετωνία ή με μια άλλη εταιρεία στη Σλοβενία, με ένα ε, πρόγραμμα ασφάλειας της μεταφοράς στην Ισπανία, με πράσινη ενέργεια για τις μεταφορές σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Μια από τις νέες εξελίξεις είναι η διευκόλυνση για την ε, διασύνδεση της Ευρώπης και τα σχετικά οι σχετικές προσπάθειες blending του συνδυασμού. Καλά έκανε η Move και η Επίτροπος Βιολέτα Μπούλτς. Τα συζητήσαμε και το πρωί. Χρειάζεται να κινητοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις προς ε, την ε, διευκόλυνση διασύνδεσης της Ευρώπης Αυτές λοιπόν οι ανακοινώσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, blending θα πρέπει να περάσουν από την ευρωπαϊκή διαδικασία για να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, εγγύησεις και να πληρώνται οι σχετικοί όροι. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε και στο μέλλον για να δούμε πώ θα καλυφθεί το χάσμα αυτό στι επενδύσει. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσω εδώ για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για ερωταπαντήσει και συζήτηση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις συζητήσεις που θα έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Χούντακ και να δώσω αμέσως το λόγο σε εσά, κύριε Βαντενκάμπ, για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. En ook de andere meneer ε, καλωσορίζουμε και τον κύριο Χούντακ από ε, την ΕΤΕΠ. Έχω μια ημιπροσωπική ερώτηση. Ε, εσείς θα αντικαταστήσετε τώρα τον κύριο Βαμπάλεκομπ ή όχι. Ε, και μπορείτε να μου το απαντήσετε πριν συνεχίσω αμέσως. Good, good question. Um, Καλή ερώτηση. Προσωρινά ε, τον αντικαθιστώ. Ξέρετε ότι ο κύριος Φαμπάλεκομ Πιμ ήταν αρμόδιος για τα θέματα των μεταφορών, αλλά δεν είναι πλέον αντιπρόεδρος είναι Οκταμελή η Επιτροπή, οκτώ αντιπρόεδροι, ο καθένας στο χαρτοφυλάκιό του και προσωρινά τώρα μέχρι να οριστεί κάποιος από την περιοχή Μπενελούξ. Έχω επιφορτιστεί εγώ με τα, των μεταφορών. Ευχαριστώ, γι' αυτό σας ρώτησα. Ήθελα να το ρωτήσω γιατί είπε ότι μπορεί να υποφέρει, ε, αλλά ας μην τον ανακρίνουμε. Όταν ο άνθρωπος σας σκέφτεται τα καθήκοντα προσωρινά, δεν χρειάζεται να τον ε, τσουρουφλήσουμε. Έχω όμως κάποιες επικριτικές ερωτήσεις. Τα 30 εκατομμύρια που αναφέρατε για επενδύσεις ε, στις μεταφορές, είπατε 17%. Τα τελευταία χρόνια αυτά δεν έχουν αυξηθεί. Μπορείτε αυτό να το επιβεβαιώσετε ή να το εξηγήσετε. Τα 30 δις όμως, που λέει τώρα ο κύριος ε, Βαντεγκάπ, ε, είναι σταθερά και δεν αυξάνονται. Τα 30 εκατομμύρια της ΕΤΕΠ, ποια σχέση έχουν με τα 25 δις εκατομμύρια ε, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι 30 συν 25. Ε, γιατί είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η σχέση των δύο ποσών μεταξύ τους. Μετά. Αυτοκινητόδρομη, σίδηροδρομη και εσωτερική ναυσιπλοεία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρειάζεται πια να επενδύσει στου αυτοκινητοδρόμους, για να το πω ε, έτσι κάπως ε, χοντρά, γιατί υπάρχουν τα διόδια αυτοκινητόδρομοι, είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι. Μήπως ε, να επικεντρωθείτε πιο πολύ στο σιδηρόδρομο και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Ήταν τρίτη ερώτηση αυτή, τέταρτη τώρα. Ξέρετε ότι εγώ είμαι Ολλανδός και οι Ολλανδικές τράπεζες σίγουρα είναι ανταγωνιστικές της ΕΤΕΠ. Νομίζω ιδιωτικέ τράπεζες είναι και πιο φθηνέ και δίνουν και πιο φθηνά επιτόκια ε, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό μπορεί να μην ισχύει σε όλε τι χώρες. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, χωρίς καμιά αμφιβολία, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πώ αντιμετωπίζετε εσείς ε, τον ανταγωνισμό με τι ιδιωτικέ τράπεζε, Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με το αφεντικό σα εδώ, ο οποίο μα είχε πει ότι Καλά, και εμείς έχουμε εμπορικές τιμές, ε, γιατί δεν είμαστε φιλανθρωπικό σωματείο και εμείς εμπορική τράπεζα είμαστε. Αλλά, εντάξει, αν στην Ολλανδία ιδιωτικέ τράπεζες μπορούν να κάνουν καλύτερες προσφορές από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μήπως χάνει το στόχο της η ΕΤΕΠ. Γιατί είναι θαυμάσιο και καταπληκτικό που κάνετε, που έχετε κέρδη δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ. Αλλά είστε Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όχι Ευρωπαϊκή Μονή Κοπή Χρήματο. Πρόεδρε, μπορεί να σα ακούγεται λίγο σοσιαλιστικό αυτό, αλλά θέλω να το στριμώξω με τι ερωτήσει μου. Μετά, τι κάνετε με το blending, αυτό το, το μείγμα χρηματοδότηση. Λέτε ότι σα αφορά και σα ενδιαφέρει. Η Γενική Διεύθυνση MOVE λέει ότι αυτοί κάνουν το blending όλο και εσείς καθόλου. Και το ίδιο για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Την αναφέρατε. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με αυτή τη διευκόλυνση. Γιατί και πάλι λέει η Γενική Κυρίευση Μόφ, αυτά τα κάνουμε εμείς. Το ΣΕΦ είναι κυρίως ε, επιδοτήσεις, έτσι δεν είναι δάνεια. Αλλά θέλω να ρωτήσω λίγα περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση της τράπεζάς σας ε, ως προς το blending και το ΣΕΦ. Και όχι οι συμβουλές, το χρήμα, το ρευστό. Ευχαριστώ κύριε Παφαντεγκάμπ. Κύριε Σίνκε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε δύο λόγια σε σχέση με δύο ακόμα ζητήματα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ξεκινούμε την ε, σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό των επόμενων ε, ετών, δηλαδή 2020-2001 ε, και μετά, από εκεί και μετά για το πλαίσιο στο 2027. Οπότε βλέπουμε ότι για την πολιτική συνοχή θα έχουμε πολύ λιγότερα κονδύλια, ενώ θα έχουμε λιγότερα κονδύλια και για τα διαφθορτικά ταμεία. Άρα λοιπόν, στον προπολογισμό της Ένωσης θα προβλέπονται ε, κατά συνέπεια, λογικά, μοιραία και λιγότερα κονδύλια για το τομέα των μεταφορών. Οπότε το ερώτημα που σα θέτω σχετικά είναι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λαμβάνει υπόψη τη αυτήν την ε, ε, μείωση στο πλαίσιο της πολιτικής παροχή δανείων της. Δεύτερο ερώτημα για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός της Ένωσης περιλαμβάνει ένα αρκετά ε, σεβαστό ε, ποσό, 6,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την κινητικότητα και σε σχέση και με την ασφάλεια και νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε με περισσότερη ευκολία διάφορε δυνάμει επιβολή τη νομοθεσία, αστυνομικέ δυνάμει και άλλε. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ανοίξει μια νέα γραμμή δανειοδότηση σε ό,τι αφορά τέτοιου είδου ε, ε, δυνατότητε αύξηση δηλαδή τη κινητικότητα και των δυνατοτήτων μεταφορά για τι αρχέ επιβολή του νόμου. Η κυρία Φώστερ δεν είναι, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι η κυρία Φώστερ. Ο κύριο Βαντάλεν όμω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Χούντακ και εγώ ε, Ολλανδός βουλευτής είμαι και στη χώρα μου διαπιστώνω μια επιφυλακτικότητα απέναντι στο ρόλο της ΕΤΕΠ. Το είπε και ο κύριος Βαντενκάμπ. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία της για ε, σχέδια και έργα μεταφορών στην Ολλανδία. Ε, γίνεται μια συζήτηση εκεί και ο κόσμος στρέφεται προς τις μεγάλες τράπεζες όπου ε, η ΕΤΕΠ απουσιάζει από τον πίνακα αυτό. Λοιπόν, σας ερωτώ, εσείς ποια προστιθέμενη αξία έρχεστε να φέρετε σε μεγάλα έργα υποδομών μεταφορών απέναντι σε άλλες μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, πολύ συγκεκριμένα. Ένα από τα έργα τα οποία συζητάμε στη χώρα μου εδώ και χρόνια είναι η ανανέωση και η μεγάλη ε, αύξηση ε, ενό υδατοφράχτη ε, στο λεγόμενο σε, σε ένα φράγμα που έχει ε, κόψει τη μεγάλη θάλασσα, την εσωτερική θάλασσα που λέγεται πέλαγος Άισελ. Ε, αυτός ο υδατοφράχτης και όλη η υποδομή έχει κατασκευαστεί στη δεκαετία του 30 και χρειάζεται ριζική ανακαίνιση. Ε, και όταν ψάχνουν χρηματοδότηση κοιτάνε προς τις Βρυξέλλες σε διάφορες ε, θέσεις του προπολογισμού, αλλά δεν ακούω κανέναν όταν αναλύει αυτό το έργο να αναφέρει τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το ξέρετε αυτό το έργο? Στο φράγμα Αυσλαντέκ, στο Άισελμερ, στο πέλαγος αυτό το ιστορικό ε, της Ολλανδίας. Υπάρχουν ε, μέσα από τον προπολογισμό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν ακούω κανέναν να αναφέρει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε να μου δώσετε καμιά συμβουλή, γιατί είμαι σε στενή επαφή με εκείνους που το έχουν αναλάβει. Δηλαδή μπορεί να μου πείτε συμπληρωματικά ότι έχετε τη δυνατότητα συγχρηματοδότηση αυτού του έργου. Να βάλετε και εσείς τα χέρια στην τσέπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τελίτσκα. thank you. just on the, on the point that is... Σας ευχαριστώ σε σχέση με αυτό το σχόλιο που έκαναν οι Ολλανδοί συνάδελφοι. Νομίζω πως είναι σαφές και για μας ε, πως το ζήτημα της προστιθέμενης αξίας δεν έχει να κάνει με το ύψος του επιτοκίου το οποίο θα παρέχεται. Ε, δηλαδή είναι πιο περίπλοκο εδώ το ζήτημα. Αλλά χωρίς να θέλω να ε, επαναλάβω το ίδιο με αυτό που ρωτήθηκε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από τη λειτουργία για παράδειγμα των χρηματοοικονομικών αγορών στις οποίες βέβαια είσαστε ένας από τους μεγαλύτερους δανειοδότες. Ε, και κατά συνέπεια έχετε και πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα. Αλλά από εκεί και μετά, αυτό που ρωτάω είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε επίπεδο χάραξη πολιτική, προκειμένου εσεί και τα, τα προϊόντα σας τα χρηματοδοτικά να γίνουν πιο ελκυστικά. Και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στο ζήτημα των επιτοκίων, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο. Ένα δεύτερο τώρα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω. Προσπάθησα ε, για ένα δευτερόλεπτο να με φανταστώ στη θέση ενός ε, πολίτη ο οποίος ε, κάθεται εδώ κάπου στις πίσω θέσεις και να σκεφτώ τι τα είχε να κερδίσει για παράδειγμα. Ε, δηλαδή, εάν επαναλαμβάνατε τα όσα είπατε συνοπτικά ε, στο ευρύ κοινό ως προς τη θέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τι θα λέγατε. Ε, γιατί εντάξει δεν θέλουμε να μα πείτε μόνο αριθμού δηλαδή ποιο είναι το ύψο των κοντιλίων τα οποία έχετε ε, ε, δώσει ω δάνεια, γιατί αυτό το έχουμε συνηθίσει από την Επιτροπή ότι έχουμε επενδύσει αυτά τα κοντιλία ή όχι, αλλά από τί και μετά πώ αξιολογείτε την χρήση αυτών των κοντιλίων, γιατί βέβαια υπάρχει πάντοτε μια αξιολόγηση των project τα οποία υλοποιούνται και έτσι είναι δυνατόν να γίνει μια ανάλυση. Οπότε, θα μπορούσατε δηλαδή να είστε σε θέση να συντάξετε μια ετήσια έκθεση που θα λέει τι ακριβώ έχει επιτευχθεί. Και σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, για παράδειγμα, αν συντάσσετε μια έκθεση, τι θα λέγατε σε ό,τι αφορά τα πραγματικά αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά τη δανειοδότηση, ε, σε ό,τι αφορά τον χρηματοδοτικό μηχανισμό, τον συνδέοντα στην Ευρώπη, το ΣΕΦ. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν την παροχή δανείων, δεν θα ήθελα ε, να αναφερόμαστε μόνο σε, με πολιτικούς όρους σε αυτό το blending και το, δηλαδή θα πρέπει κανείς να συμμετάσχει ή όχι. Γιατί νομίζω θα πρέπει να ε, εξετάσουμε εδώ όλα τα, τα, τα διάφορα συστήματα, δηλαδή ε, σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ιδιωτική χρηματοδότηση από ιδιωτικούς επενδυτές. Εάν δούμε λοιπόν όλο αυτό, το, άλλο αυτή την εικόνα, πώς θα δούμε το πράγμα. Γιατί αν είμαι εγώ για παράδειγμα ιδιωτική τράπεζα, αν κάτι πάει λάθος θα θέλω να επαναπτύξω πατρίσω τα χρήματά μου. Οπότε ε, όταν γίνει κάτι τέτοιο, όταν υπάρξει μια κατάρρευση για παράδειγμα, αν αποτύχει κάτι, πώς θα μείνομαστε από κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι θα θεωρούσατε εσείς ως τα καταλληλότερα εργαλεία για την ε, χρήση του blending. Γιατί θα ήθελα βέβαια το blending να οδηγήσει τελικά σε μια βελτίωση του συνδυασμού των δυνάμεων σε αυτό το σύστημα. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα σημεία συμφόρηση εντό εισαγωνικών στο πλαίσιο του blending και ποιο ε, ε, θα ήταν ο καλύτερο τρόπο ή τα καλύτερα στοιχεία για να συμπεριλάβουμε σε μια μελλοντική νομοθεσία για το blending. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταλόνα. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Χούντακ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι κάποια προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν και ως ε, φιλικά για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές, φιλικά προς το περιβάλλον, τελικά δεν ήταν έτσι. Για παράδειγμα, ε, η διασύνδεση της Μπρατισλάβας ε, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕΠ με όλες τις δυνατότητες ε, των φιλικών προς το περιβάλλον και για την αντιμετώπιση των ε, κλιματικών αλλαγών. Υποτίθεται ότι θα παρότρινα τους ανθρώπους αυτούς ο περιφερειακός να περάσουν από τη χρήση των γιοταχή στις ε, συγκοινωνίες. Επίσης, υποστηρίξατε τους αυτοκινητοδρόμους μέσα των συμπράξεων ιδιωτικού δημόσιου τομέα Και δεν ξέρω κατά πόσον έχετε λάβει υπόψη τα πανευρωπαϊκά δίκτυα βάση και τη Συμφωνία των Παρισίων. Τα Υπουργεία λοιπόν που γνωρίζουν τα, των, τον ε, του ΕΦΣΥ με την εξάρτητα επιλεξιμότητα, ερεσιμότητα πώς θα μπορέσουν να λάβουν χρηματοδότηση για προγράμματα και πώς θα λαμβάνει αυτή υπόψη της ΕΤΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταλούντε. Κύριε Ρικέ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω πέντε ερωτήσεις. Η πρώτη είναι και ερώτηση και παρατήρηση. Ο ίδιος ο μηχανισμός του F.C. εν προκειμένου αυτό το κομμάτι που βρίσκεται εντός της ΕΤΕΠ, υποτίθεται ότι θα έδινε ποιοτική ε, έμφαση στην ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και όχι στα της αγοράς. Γιατί θεωρείται ότι τα προγράμματα που επιλέγονται έχουν και προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία υποτίθεται. Δεύτερη ερώτηση για την εγγύηση της πρώτης απώλειας, πράγμα που είναι μέρος του μηχανισμού και καταγράφεται και στη σύμβαση με την ΕΤΕΠ συνήθω. Όμω, βλέποντα τι συμβάσει που υπογράψατε για, τα πρώτα, για την πρώτη φάση των κοντελίων τη σηματοδότηση, δεν φαίνεται να καλύπτεται η εγγύηση αυτή τη πρώτη απώλεια. Την ανέλευαν τρίτη συμβαλόμενη, κάτι που είναι τελείω αντίθετο με το ίδιο το πνεύμα του ΕΦΣΥ. Διότι η αρχή που ε, ισχύει είναι ότι αν μειωθεί αυτό το ποσοστό του κινδύνου από εμά, τότε κινητοποιεί το ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν να αισθάνονται καλυμμένοι ως προ τον κίνδυνο. Στην περίπτωση λοιπόν που ε, κινητοποιεί, κινητοποιήσετε εσείς πώς ε, θεωρείτε ότι υπάρχει εξασφάλιση από τον κίνδυνο της πρώτης απώλειας. Και από την άποψη τη λογιστική, μετά από τρία χρόνια, τι γίνεται με το Ταμείο των Εγγυήσεων. Εάν μπορείτε να μα το πείτε βέβαια. Δηλαδή τα ποσά που καταβλήθηκαν για να υπάρχει πόσο εγγύσεων. Κάποια δι στην αρχή, 221 ε, δι στην αρχή. Ποιο είναι το κομμάτι αυτό που έχετε ε, διατηρήσει και τι έγινε με τις πρώτες επιστροφές. Πήγαν τα ποσά εκεί που έπρεπε, είναι πολύ νωρί για να μας το πείτε. Όμω μετά από τρία χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιε πρώτε επιστροφέ. Διότι υπάρχει και μια ορίμανση μετά από μια διετία για τα περισσότερα από τα έργα. Και Τέταρτη και προτελευταία ερώτηση. Η Επιτροπή που λαμβάνει τις αποφάσεις για τις κλασικές δραστηριότητες της τράπεζας, η Επιτροπή αυτή για τις ε, δεσμεύσεις σε σχέση με το ΕΦΣΙ, είναι η ίδια με αυτήν που λαμβάνει τις αποφάσεις για τις κλασικές ε, δράσεις της τράπεζας και αν όχι, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτής της Επιτροπής του ΕΦΣΙ για να υπάρχει και συνέπεια με τον ε, ίδιο το μηχανισμό. Και μια τελευταία σύντομη ερώτηση που συμπληρώνει αυτή του σοσιαλιστή συναδέλφου. Δεδομένου του καταστατικού της ΕΤΕΠ, δεν μπορείτε να παρεύετε στον τομέα της άμυνας. Ποια θα είναι όμως η θέση σας για τα 6,5 δις του δεύτερου μέρους της ε, διευκόλυνσης της διασύνδεσης της Ευρώπης. Υπάρχουν κάποιες υποδομές που είναι μικτές ας πούμε, και θα έπρεπε να καλύπτονται από αυτά τα επιπλέον ποσά για τα 6,5 δις. Δεν θα επιτρέψετε καμία κινητοποίηση γιατί υπάρχει κάποια αυτή στιγμή τόσο η αμυντική ή θα καλύψετε εσείς την ε, διάσταση της συνιστός αυτή την πολιτική, αυτή που δεν είναι αμυντική. Κύριε Ρικέ, πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Χούντακ. Αλλά κύριε Χούντακ, σας δίνω το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ε, βλέπω ότι το πνεύμα είναι καλό. Ε, μου θυμίζει κάπως τις Εθνικές Βουλές. Αλλά ελπίζω ότι και για την ΕΤΕΠ θα τα πάμε καλά ως προς την ενημέρωση και στο μέλλον. Και από το συνάδελφο που ασχολείται με τα θέματα των μεταφορών ειδικά θα ζητήσω να συμπληρώσει μετά ε, για να απαντήσει κάποιες από τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με αυτή που μου φαίνεται ότι απηχείται και στις ερωτήσεις σας σε κάποια στιγμή, το θέμα της προσθετικότητας. Η ΕΤΕΠ έρχεται να προσθεθεί σε κάτι άλλο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι ανταγωνιστική προς τους ε, δανειοδότες της, των εμπορικών τραπεζών. Ποια είναι η αξία της τα έργα γενικώ. Τι προσφέρει. Και επειδή τώρα οι συνθήκες οικονομικέ οικονομικές είναι καλές στην Ευρώπη και τα επιτόκια ε, είναι χαμηλά, ποιος είναι ο ρόλος της ΕΤΕΠ σχετικά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω βάσει της δικής μου εμπειρίας, γιατί ήμουν και σε εμπορική τράπεζα 16 χρόνια πριν αναλάβω στην κυβέρνησή μας. Ξέρω από εμπορικέ τράπεζες. Ε, πιστεύω και πραγματικά ακόμα το ε, επεξεργαζόμαστε τη συνιστόσα τη προστατικότητας στην τράπεζα για να βρούμε το σωστό δρόμο. Αλλά χρήσιμο θα ήταν να είσαστε σε μια συνάντηση τη διαχειριστική επιτροπή. Αν ήσασταν εκεί ω Ευρωβουλευτέ, για να δείτε πόσε ερωτήσει υπάρχουν πάντοτε για, κάποια, για κάθε έργο σε σχέση με την προστατικότητα. Είναι σημαντικό κριτήριο και το χρησιμοποιούμε πάντοτε για την επιλογή των προγραμμάτων. Μια από τι σημαντικότερε διαστάσει αν οποιοδήποτε έργο που εγκρίθηκε από την ΕΤΕΠ, όχι μόνο μέσω του ΕΦΣΥ, αλλά και ασχέτως, ε, δεν μπορεί παρά να έχει ένα λεγόμενο marking up. Αυτό γιατί το έργο μπορεί να έχει ψηλότερο κίνδυνο ή ξεπερνά τα σύνορα του ενός κράτους, έχει ευρωπαϊκή διάσταση, άρα είναι πιο δύσκολο να το αναλάβει ένα κράτος. Ή υπάρχουν άλλα θέματα που άπτονται του κενού στη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου. Ας πούμε, η κοινωνική στέγαση. Κάτι σχετικό υπάρχει και στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Ε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ε, εμπορικές τράπεζες να δώσουν δάνεια σε αυτόν τον αλλά υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να δώσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τότε οι εμπορικέ τράπεζε μπορούν να πάρουν τα επιτόκια που έχει και η ΕΤΕΠ, αλλά για συντομότερο διάστημα. Δηλαδή μπορούν να χρηματοδοτήσουν για 7 χρόνια περίπου η ΕΤΕΠ, χάρη στο γεγονό ότι έχουμε τριπλό Α στις διεθνείς αγορές και είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρήματα που χρησιμοποιούμε είναι ποσά ε, επενδυτικών ταμείων, συνταξιδοτικών. Ένα τρίτο έρχεται και από τη ΣΥΠΑ. Έχουμε λοιπόν και την εμπορική μας ε, διάσταση. Χάρη σε αυτήν την ε, διάσταση μπορούμε να δώσουμε διάρκεια και 20-25 χρόνια στα δάνεια μεγάλη ορίμανση. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τους περισσότερους ε, δανειοδότες του εμπορικού ε, τομέα. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το μακρύτερο διάστημα χρηματοδότησης σε σχέση με τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά τα άλλα, χρηματοδοτούμε περίπου 50% του έργου πολύ. Άρα χρειαζόμαστε και κάποιον εταίρο οπωσδήποτε. Επενδυτικό ταμείο, επενδυτοπορική τράπεζα, εθνικά ή περιφερειακά κονδύλια ε, για να έρθουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αλλιώς το έργο δεν θα εκτελεστεί. Αυτό είναι μέρος των προποθέσεων για οποιοδήποτε έργο για το οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από το 50% της χρηματοδότησής του. Με το ΕΦΣΙ βεβαίω υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Το ΕΦΣΙ 2, α πούμε, που είναι μέρο τη εξίσωση για την υποστατικότητα. Υπάρχει και η Επιτροπή Επενδύσεων. Ναι, το ΕΦΣΥ βασίζεται στην υπόθεση ότι θα καλυφθούν έργα που έχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου. Έργα που η ΕΤΕΠ δεν θα υποστήριζε αλλιώ. Ούτε εμπορικές τράπεζες δεν υποστήριζαν. Θυμάμαι ακόμη τι έλεγαν οι Υπουργοί Οικονομικών το 2013 σε μια συνεδρία σε Κοφίν και έγινε μια συζήτηση, νομίζω έλεγαν ο Σόιμπλε και άλλοι, γιατί πρέπει να υπάρξει ποσοτική χαλάρωση και η ΕΚΤ ε, χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να υπάρξει ρευστότητα στι αγορέ. Και δεν βλέπαμε να χρηματοδοτούνται έργα στην πραγματική οικονομία. Πολλοί υπουργοί συμφώνησαν τότε ότι ένα από του λόγου ήταν το υψηλό επίπεδο κινδύνου για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων και ότι αυτό πρέπει κάπω να καλύπτεται. Επίσης, οι εμπορικές τράπεζες, λόγω της οικονομικής κρίσης, ε, είχαν τόση ρύθμιση, τόσους κανόνες να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα προς τα προς την κεφαλαιοχική του σύσταση και ούτω καθεξής. Οπότε το ΕΦΣΥ έδωσε τις εγγυήσεις, ε, με τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΤΕΠ για να καλυφθεί αυτή η διάσταση του κινδύνου. Όμως σε σχέση με την απόφαση για τις εγγυήσεις και ποιο έργο θα πάρει εγγύηση από το ΕΦΣΥ, αυτό αυτή την απόφαση τη λαμβάνει ανεξάρτητο φορέα, η Επιτροπή Επενδύσεων. Και στο FC2 το είχαν ζητήσει και οι ευρωβουλευτέ. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε που αποφασίζουν εκτός του management της ΕΤΕΠ ποιο έργο ε, μπορεί να πάρει ε, εγγύηση. Και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό έργων που, έχει υποστηριχθεί, ε, το, ως το, που έχουν υποστηριχθεί ως τώρα από το ΕΦΣΥ που είχαν ποσοστό κινδύνου δίμιον έργα που σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί από κανονικές προσπάθειες χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια αυστηρότατη διαδικασία διασφάλιση ότι κάθε έργο που, προσ... χρηματοδοτεί η ΕΤΕΠ διαθέτει αυτήν την προσθετικότητα. Υπάρχει αυτό το κενό της αγοράς, όπως το λέμε, το market gap, για την ε, επιλογή τέτοιων έργων. Τώρα για τους ε, συγκεκριμένους αριθμούς που ρώτησε ο κύριος Κάμπ, το 17% ε, της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ, τα 13 δις αύξηση, τα 25 δις ε, μόχλευσης. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο να τα πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Να προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικές από τις λεπτομε... επιμέρους ερωτήσεις που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Βαντεγκάμπ. 13 ήταν ο αριθμό, 13 όχι 30, 13 δι. Θα θέλαμε να είναι 30. Σε κάθε περίπτωση όμως θέσατε την ερώτηση αν το ΕΦΣΙ και τα 25 δις έρχονται να προσθεθούν στα 13. Καλή ερώτηση, απάντηση είναι όχι. Η εγγύηση του ΕΦΣΙ λειτουργεί με περισσότερη μόχλευση από ότι αυτά που κάνει συνήθω η ΤΕΠ. Τα 25 δις βασίζονται στο 1 δεκατοπέμπτο των πραγματικών κονδυλίων που παίρνει η τραπεζα. Υπάρχει ένας λόγος 1 προς 15 για τη μόχλευση των έργων του ΕΨΗ. Και αυτό γιατί το κρατικό χρήμα ε, φέρνει, κινητοποιεί περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια. Ε, οι κανονικές δραστηριότητε τη ΕΤΕΠ και το είπε και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πάνω από 50% ενός έργου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, χρηματοδοτούμε πολύ λιγότερο. Κατά μέσο όρο είμαστε στο 3 έω 4% ω πολλαπλασιαστής. Εάν ε, χρηματοδοτήσουμε 100 εκατομμύρια, εάν δανείσουμε 100 εκατομμύρια, φτάνουμε τα 150 στι επενδύσεις συνολικά. Αυτή είναι η δική μας προστιθέμενη αξία. Εδώ έχουμε προγράμματα διαφόρων ειδών χρηματοδότηση και όπω είπαμε και με την ε, εμπλοκή του δημόσιου και με τη συμπράξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στηρίζουμε όλα αυτά τα είδη προγραμμάτων και έργων, αλλά η επιλογή της χρηματοδότησης πολλές φορές είναι θέμα των κατών μελών και του συγκεκριμένου ανάδοχου. Δεν τον επιλέγουμε εμεί. Απλώ κοιτάζουμε το είδο χρηματοδότηση, βεβαιωνόμαστε ότι είναι ευρωπαϊκό το έργο, ότι οικονομικός μπορεί να είναι αποδοτικό και ότι συμφωνεί με, τις, ε, με τους κανόνες της δανειοδότησης που ακολουθούν και όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική. Νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος απάντησε κάπως το ερώτημα για τι ε, τράπεζε, τι Ολλανδικέ τράπεζε οι οποίε μπορούν να πάρουν δάνεια φτηνά στι αγορέ σχετικά και υπάρχουν, είμαστε στι συνθήκε τη αγορά. Υπάρχουν κομμάτια του κλάδου των μεταφορών, υπάρχουν ε, πράγματα στην Ευρώπη που δεν είναι ελκυστικά στου επενδυτέ. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να πάρει τα χρήματά μα. Οπότε εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που έχουμε για τα έργα. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια επιπλέον ε, ε, αξία στα έργα που να φέρει τους επενδυτές και τους αγοραστές. Πάντως το έργο που αναφέρατε θα ήταν οπωσδήποτε επιλέξιμο. Αλλά θα μπορούσαν νομίζω και οι ίδιοι να πάρουν ευθυνά δάνεια για να το χρηματοδοτήσουν. Ε, τον κύριο Ζέμ και το ερώτημα που έθεσα, σα ευχαριστώ. Ε, θέσατε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πολιτισμικό δημοσιονομικό πλαίσιο και την ε, πρόταση για περικοπέ ε, που έγινε από την πλευρά τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική συνοχή, δηλαδή τα σχετικά κοντήλα και τι αυτό θα σήμαινε για την πολιτική μεταφορά αλλά και για το δικό μα ρόλο ω ΕΤΕΠ. Ε, θεωρούμε πως αυτή η μείωση της χρηματοδότησης ε, για την πολιτική συνοχή αποτελεί, ε, αν θέλετε, φυσική συνέπεια του Brexit, της νέας δηλαδή δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά και του γεγονότο διαφορετική κατάσταση ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που αποφελούνται από την πολιτική συνοχή. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι δίκαιο ή όχι να συμβαίνει. Πάντω, εμεί δραστηριοποιούμαστε σε δύο κυρίου τομεί. όπως έχει ήδη καταδείξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, ε, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια και ε, του ε, προϋπολογισμού προκειμένου να κινητοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια και άλλα είδη χρηματοδότησης μέσω δηλαδή της όθησης που δίνουν. Για παράδειγμα, μέσω του ΕΦΣΥ με 21 μόνο δισεκατομμύρια μπορούμε ε, να προσελκύσουμε 315 δισεκατομμύρια, δηλαδή να μοχλεύσουμε με αυτόν τον τρόπο άλλα κεφάλαια, με την όθηση που δίνουμε ένα αρχικό κεφάλαιο μέσω αυτών των κοντιλίων. Και νομίζω αυτό είναι ένα ε, τρόπο που καταδεικνύει πώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον έργα τη ε, πολιτική συνοχή. Άρα λοιπόν, εμεί από την πλευρά τη ΕΤΕΠ και με βάση την εμπειρία που έχουμε από το ΕΦΣΙ θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη αξιο, ε, αξιοποίηση των ε, ε, χρηματοδοτικών εργαλείων, έτσι ακριβώς να κινητοποιήσουμε, να απομοχλεύσουμε ιδιωτικά κονδύλια. Και βέβαια αυτά τα, με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν τα συνολικά κονδύλια που επενδύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν θα προσελκύσουμε περισσότερα επενδυτικά κονδύλια και στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η τεχνική αρρωγή που παρέχουμε. Δηλαδή ε, το να αναπτύξει κανείς ένα project το οποίο μπορεί να έχει μια τέτοια επίδοση δεν είναι εύκολο. Και στις χώρες που αποφελούνται από την πολιτική συνοχή, οι αρχέ τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση αλλά και ε, οι επιχειρηματίε ε, κατά κάποιο τρόπο είναι εθισμένοι εντό εισαγωγικών σε ενισχύσει, σε άμεσε επιδοτήσει, δηλαδή σε δωρεάν εντό εισαγωγικών χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, άλλα project τα οποία ε, ε, κατά το ένα μέρος τους θα πρέπει βέβαια να επαναχρηματοδοτούνται πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει και έτσι λοιπόν εμείς από το δικό μας τρόπο υποστηρίζουμε τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες όπως την EGK για παράδειγμα και άλλες στην Πολωνία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη προκειμένου αυτές οι τράπεζες να αναπτύξουν αν θέλετε μια νέα νοοτροπία αλλά και τις κατάλληλες δεξιότητες για να διαχειρίζονται τέτοια νέα έργα. Ε, και εμείς από την πλευρά της ΕΤΕΠ θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρέχουμε αυτή τη τεχνική ε, ε, βοήθεια προκειμένου να επιτρέψουμε και στους δικαιούχους σε αυτές τις χώρες της πολιτικής συνοχής να αναπτύσσουν νέου είδους προγράμματα αν θέλετε. Τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κινητικότητας και της ασφάλειας, δηλαδή των σχετικών αρχών ασφαλείας, Είχαμε τη συζήτηση σήμερα με τον Επίτροπο Πούρση και έγινε μια αναφορά σε μια νέα πρωτοβουλία με τον με την ονομασία ε, ασφάλεια στι οδικέ μεταφορέ, γιατί πραγματικά παραμένει ε, υψηλό ο αριθμό των ε, θυμάτων ε, τέτοιων αυτοκινηστικών ε, ατυχημάτων. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα όλε τι επιμέρου παραμέτρου, έτσι ώστε οι δρόμοι μα να γίνουν και ασφαλέστεροι για του ανθρώπου μα, αλλά και καθαρότεροι για το περιβάλλον. Και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε μια νέα κοινή πρωτοβουλία ΕΤΕΠ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια ε, στο δρόμο, αλλά προκειμένου να αυξήσουμε και την κινητικότητα των ανθρώπων εντό των κρατών μελών του αλλά και διασυνοριακά. Αντιπρόεδρε Τέλεσκα, απαντώντας σε αυτό που είπατε, Δηλαδή το πώς, ε, πώς είμαστε ελκυστικοί ως ΕΤΕ πέραν των επιτοκίων που χορηγούμε. Ε, ένας από τους τρόπους που μπορούμε να το επιτύχουμε, αυτό που μας διαφοροποιεί αν θέλετε από τις εμπορικές τράπεζες, είναι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ε, που παρέχουμε και η οποία γενικότερα δεν είναι διαθέσιμη από τις εμπορικές τράπεζες. όπως θα γνωρίζετε, είμαστε για παράδειγμα αυτή την περίοδο σε διαβούλευση με, την με το Συνδρομικό Οργανισμό της ε, Τσεχίας σε ό,τι αφορά μια νέα χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τι 4 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο δίκτυο το συνδρομικό στην Τσεχία και αυτό βέβαια ε, δίδεται ως χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και, από, και όχι από ιδιωτικέ ε, τράπεζες γιατί ακριβώ μπορούμε να παράσχουμε βάθο χρόνου σε χρηματοδότηση 20-25 ετών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο επιτρέπει ακριβώ την ε, την διέρεση αν θέλετε τη ε, της επαναπληρωμής ε, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κάτι ακόμα τώρα που μπορεί να παράσει περισσότερη προμεστηθέμενη αξία είναι η η δυνατότητα που έχουμε να διαστρώνουμε καλύτερα τα προγράμματα και να συνδέουμε καλύτερα την καινοτομία με την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, στην Τσεχία και γενικότερα σε χώρε τη Κεντρική Ευρώπη που αποφελούνται από το καδουλία συνεχή, έχουμε αυτή τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τι έξυπνε πόλει και τι έξυπνε περιφέρειε, smart cities, smart regions σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε project τα οποία έχουν και μια πτυχή καινοτομία σε τοπικό επίπεδο. Και εδώ εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε μάλλον και, και με την ε, Τσεχική ε, ε, Τράπεζα για την, αυτή την περιφερειακή ανάπτυξη ακριβώς στο πλαίσιο τέτοιων project. Και, και σε αυτό το τομέα οι εμπορικές τράπεζες δεν είναι έτοιμες να παράσχουν μια υποστήριξη έτσι όπως την παρέχουμε εμείς δηλαδή με φτηνή χρηματοδότηση, με τεχνική υποστήριξη, με τη σωστή συνοχή και τη σωστή διάρθρωση των προγραμμάτων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προσφέρονται από τις εμπορικέ τράπεζες. σε ό,τι αφορά τώρα το blending, τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο ειδικότερα του ε, ΣΕΦ και τα σημεία συμφόρηση, αν θέλετε, στο πλαίσιο αυτή τη χρηματοδότηση του blending. Και για μα να πούμε ότι πρόκειται για μια νέα εμπειρία εδώ. Δηλαδή αυτό το blending του ΣΕΦ. Και ίσω ο Γκάβιν μπορεί να, πει περισσότερα σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά ε, κατά τη δική μας άποψη εκείνο που είναι το βασικό πρόβλημα είναι τα project τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη τέτοιων ε, project. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιου είδου ε, project, αλλά πραγματικά πολύ λίγα από αυτά στον χώρο των μεταφορών είναι πραγματικά χρηματοδοτήσιμα. Δηλαδή ε, πολλέ ε, αρχέ τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πολλέ κυβερνήσει θεωρούν πω μπορούν απλώ να κάνουν μια μετάβαση από, το, από την ενίσχυση, την άμεση, στο blending. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, αν κανεί θέλει να παράσχει blending, θα πρέπει να υπάρχει και ένα ε, ζήτημα απόδοση, ε, μια πτυχή απόδοση αυτού του project υπό οικονομικού όρου. Οπότε ε, βρισκόμαστε ε, αυτή την περίοδο σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώ μπορεί αυτό να, ε, να βελτιωθεί στο μόνο, δηλαδή σίγουρα θα χρειαστεί εδώ περισσότερη ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χοντάκ. Μπορούμε να το χειροκροτήσουμε φυσικά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μας πείτε συγκεκριμένα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έλα, αυτό το ερώτημα ε, παρέμεινε αναπάντητο. Ο κύριος Νταλούντε ε, ρώτησε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση και τη χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ. Εσείς χρηματοδοτείτε αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα. Πώς θα επιλέγετε, με ποια κριτήρια. Ε, ποια είναι τα κριτήρια λοιπόν. Και ο κύριος Ζεκέ έκανε πέντε ερωτήσεις, δεν απαντήσατε. Να σας ξαναδώσω το λόγο πολύ σύντομα. Και ο κύριος Δαλούντε, ναι. Μήπως θέλετε να απαντήσετε, ναι. Α, ο συνάδελφός σας, καλώς. Ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια μόνο για την κλιματική δράση και την επιλογή των έργων. Βεβαίως, επενδύουμε ε, σε όλο το φάσμα και σε όλους τους τομείς των μεταφορών και όλα τα μέσα μεταφορών. 25% είναι ο στόχος μας ε, για τη δανειοδότηση των μεταφορών και όλη τη δανειοδότηση να ε, ταξινομηθεί ως ενέργεια για την προστασία του κλίματος, για το μετριασμό, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εξάντε, εκ των προτέρων δηλαδή, ε, επιλέγουμε αυτά τα έργα για να ανταποκριθούμε στους στόχους ε, της προστασίας του κλίματος. Ε, στις μεταφορές τι γίνεται. Η δανειοδότησή μας είναι προς το σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και σε κάποιο βαθμό λιμένες και κυρίως περιαστικούς σιδηροδρόμους αλλά και αστικούς σιδηροδρόμους. Είναι πολύ σημαντικές οι πόλεις για μας, ε, για τη δραστηριότητά μας και το θεματολόγιο το, της διασύνδεσης των πόλεων, ας πούμε καλύτερα συστήματα μετρό ε, και τραμ σταθερής τροχιάς ε, στις αστικές περιοχές. 60% λοιπόν περίπου του δανεισμού μας πηγαίνει προς ε, την κατεύθυνση αυτή, στις μεταφορές, προς πιο αηφόρες μορφές και μέσα μεταφορών. Και σε ό,τι αφορά τη συνολική δανειοδότηση έχουμε στόχο 25% υπέρ των κλιματικών δράσεων που τον επιτυγχάνουμε κάθε χρόνο. Και ρωτήσω του κύριου Ρικέ. Α, να απαντήσω και σε αυτές και στις 5. So I think if I have it correctly... Εάν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε για το ΕΦΣΙ και την προστιθέμενη αξία του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε αυτό απάντησε νομίζω ο Αντιπρόεδρος. Για τους τομείς τώρα που είναι ζημιογόνοι και που χάσαμε χρήματα, εξ γνωρίζω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που να καταφύγουμε στην εγγύηση. Αυτό θεωρείται κανονικά θετικό. Θα δούμε στην πορεία των έργων αν θα παραμείνει. το σημαντικό είναι ότι υπάρχει εγγύηση σε περίπτωση που χρειαστεί για να μπορέσει να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Για τις επιστροφές από τις εγγύησεις που έχουν καταβάλει τα κράτη-μέλη, τι εννοείται ακριβώς. Ε, ε, ε, έχει σχέση με το εισόδημα αυτό και με το, το ποσό Έχουμε μια ε, μόχλευση 15 ε, 15 πλάσια δηλαδή της αρχικής από τα 21 δις έγιναν 315 σε γνωρίζω δεν έχουν γίνει υπολογισμοί για το, τη χρηματική αξία αυτών in Καλά, μπορεί να είναι ζημιογόνα υπό μία έννοια αυτή η ε, δράση. Η ερώτηση για την Επιτροπή Εύση του Ταμιστοτήκων Επενδύσεων νομίζω έχει απαντηθεί. Α, μια πολύ καλή ερώτηση που δεν ε, εξετάσαμε ακόμα. Είναι το θέμα της άμυνας. Uh, ε, ουσιαστικά ο πρόεδρος ε, της τράπεζας, ο κύριος Χόιερ, είχε ανακοινώσει πριν από ένα χρόνο περίπου ότι η τράπεζα λανσάρει μια δική της πρωτοβουλία για την ασφάλεια Έχω ξεχάσει τα ακριβή ποσά, δύο δις νομίζω, επενδύσεων ε, που θα υποστήριζε η τράπεζα και θα συμμετείχε, ε, επενδύσεις έργα σχετικά με την ασφάλεια. Και ε, εκεί έχουμε και έργα και επενδύσεις υποδομές διτής χρήσης, στρατιωτικής και πολιτικής. Αυτό αναφέρεται σε νέα πρωτοβουλία. Η απάντηση είναι ότι η τράπεζα έχει ήδη λάβει θέση. Ότι διτή χρήση σημαίνει ότι μπορούμε να συμμετέχουμε ως προς το πολιτικό σκέλος. Αυτό μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας, εφόσον υπάρχει τέτοιο πολιτικό σκέλος και ε, έχουμε την πρόθεση να ε, επενδύουμε δύο δις ετησίως στην κατεύθυνση αυτή, σε έργα διτής χρήσης. Ο κύριος Βαντενκάμπ ζητεί το λόγο. Έχουμε ακόμα 8 λεπτά. Και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, οπότε με φιδώ το χρόνο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά τα 13 λοιπόν δισεκατομμύρια, γιατί έχω μπερδευτεί. Αυτό είναι για το 2017, για μεγαλύτερη περίοδο γιατί το έχω χάσει λίγο. Οι επενδύσεις τη ευρωπαικη Τράπεζας επενδύσεων 13 δις, Ετησίω. Ετησίω, μάλιστα. Πρόεδρε, γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει και σας πάρα πολύ το θέμα αυτό. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εσεί, μιλήσατε για ασφάλεια, security. Εμεί μιλήσαμε για άμυνα, για στρατιωτικέ παύλα, αμυντικές μεταφορέ. Δηλαδή, αν κάνει καλύτερα ε, κανένα στη φύλαξη των αεροδρομίων ε, με χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για καλύτερη φύλαξη, αυτό είναι ασφάλεια, αλλά δεν είναι άμυνα όταν έχετε συστήματα, ας πούμε, με έλεγχο των διόδων και τα λοιπά. Εσείς κάνετε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στην άμυνα και την ασφάλεια. Εξηγήστε το παρακαλώ. Ε, ορίστε, έχετε το λόγο, κύριος Χούντακ. Όπως σας εξήγησα, εμείς είμαστε τράπεζα δημόσια, αλλά χρησιμοποιούμε και πόρους από ε, ιδιωτικά ε, ιδρύματα, hedge funds, συνταξιδοτικά ταμεία κλπ. Ε, Παγκοσμίω. Και μεταξύ των επενδυτών υπάρχουν κάποιοι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την άμυνα, σε οτιδήποτε μπορεί να χρηματοδοτήσει όπλα που σκοτώνουν κλπ. Όταν λοιπόν καλούμαστε να ορίσουμε το ρόλο μας ε, στο χώρο της άμυνας και της ασφάλειας, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι που θα πάμε προς την αμυντική βιομηχανία χωρίς να χάσουμε κάποιους σημαντικούς επενδυτές ε, από τα ομόλογά μας. Αυτό είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Ε, για την ασφάλεια μιλούμε και για τεχνολογίες και έργα της χρήσης, όπου υπάρχει και ένα ισχυρό πολιτικό σκέλος και όχι μόνο αμυντικό ή στρατιωτικό. Και η κυβερνοασφάλεια επίσης, που γνωρίζουμε ότι στη σύγχρονη άμυνα είναι όλο και πιο σημαντική και δεν είναι ε, τα παραδοσιακά άρματα μάχης και ο βαρύς ε, οπλισμός, αλλά είναι πιο περίπλοκες αμυντικοί που δράσεις. Εκεί θέλουμε και έχουμε την πρόθεση να δραστηριοποιούμαστε. με ελάχιστη συμμετοχή 2 δισεκατομμύρια ετησίω. Ευχαριστώ. Είχα και εγώ μια ερωτησούλα τελευταία, πάρα πολύ μικρή όμω. Τι είδαμε στο Dieselgate, υπάρχουν κατασκευαστές αυτοκινήτων που χρησιμοποίησαν τα δάνεια ε, της ΕΤΕΠ ως μη όφυλαν. Και πολύ ε, συγκεκριμένη και απλή ερώτηση. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα θεσπίστε έτσι ώστε τα δάνειά σας δεν βοηθούν τους κατασκευαστέ αυτοκινήτων να κάνουν ό,τι να είναι. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανετικές συνέπειες ε, με την ρήπαση, την ατμοσφαιρική και τα αέρια του θερμοκηπίου. Um, okay. I mean, our, our supports... Η υποστηρίξή μας προς την αυτοκινητοβιομηχανία και τη, τα, βιομηχανία των οχημάτων οδικών μεταφορών είναι ω προ την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Κατά κύριο λόγο. Αυτέ οι τεχνολογίε που αναπτύχθηκαν είχαν ε, διαδοθεί ευρέω. Ε, αυτό είναι ένα από τα χάσματα όμω τη αγορά που με χαρά να έρθουμε να καλύψουμε. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλε προηγμένε βιομηχανικέ οικονομίες. Ω προ την έρευνα και την καινοτομία και την ανάπτυξη. Η βασική μας λοιπόν συλλογιστική θα είναι αυτή. Μετά υπάρχει και το θέμα το ότι έχουμε έναν ή δυο πελάτες οι οποίοι μας εξαπατούν. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό βεβαίως εφόσον ανοιχτηθεί με τη δέουσα επιμέλεια και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλέσουμε κάποιες σηματοδοτήσεις. Τώρα αυτού του είδους η απάτη εντό εισαγωγικών έχει εντοπιστεί και βεβαίως βάσει της κλασικής μας δραστηριότητα και χάρη στους εμπειρογνωμονές μας έχουμε το νου μα για τέτοιες περιπτώσεις. Η καλύτερη διασφάλιση για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον είναι αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Αισθανόμαστε όλοι μεγάλη ανακούφιση λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Χούντακ. Και που μας αφιερώσατε χρόνο για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της ΕΤΕΠ και το τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, τι προκλήσεις. Μόλις είχαμε μια συζήτηση με τον εισηγητή μας, ε, κύριο Τέλιτσκα, για τις μεγάλες προκλήσεις του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Εδώ, αυτό που μας ενδιαφέρει ως προς το έύση, γιατί το συζητήσαμε διαμακρόν εδώ, είναι τι γίνεται με τη διασύνδεση. Και αν δούμε το σύνολο των έργων που χρηματοδοτούνται, 9% μόνο αφορούν τι μεταφορέ. Θα πρέπει να υπάρξει πολλαπλασιασμό επί 2, επί 3 και επί 4 για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που μόλι έχουμε περιγράψει και που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, μπορείτε να τον χειροκροτήσετε. Allez, nous continuons nos travaux. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στη συγγήτριά μα την κυρία Γιώτο και καλημέρα σα. Ε, θέμα. Κοινοί κανόνε για ορισμένε συνδυασμένε εμπορευματικέ μεταφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Έχετε το λόγο, κυρία Γιώτο μου, και μετά οι διάφοροι σκιώδη εισηγητέ. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος της Κομισιόν. Εσείς κυρία Κοσέτσκα θα πάρετε το λόγο. Ωραία λοιπόν. Ακούσουμε πρώτα την εισηγητριά μας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές, διότι πραγματικά η δουλειά που κάναμε ήταν φανταστική και σίγουρα αποτελεσματική. Πιστεύω ότι θα οδηγήσουμε σε αίσιο πέρα στο όλο θέμα, δεδομένων όσων έγιναν τώρα. Η κοινή μας δουλειά μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μία πρόταση που κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά σωστά εξισορροπημένη, διότι λαμβάνει υπόψη τα περισσότερα από τα αιτήματα που έθεσαν και οι άλλες ομάδες. Στη δική μου αρχική πρόταση είχα συμπεριλάβει μια σειρά από μέτρα με σκοπό να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους συνδυασμένου τρόπους μεταφορών, τους διατροπικούς, για να καλυφθεί αυτό το gap, αυτό το χάσμα μεταξύ των εντό εισαγωγικών κλασικών αποκλειστικών μεταφορών σε σχέση με τις συνδυασμένε. Και αυτό γιατί σήμερα οι διατροπικές μεταφορές ε, χρησιμοποιούνται με ποσοστά πραγματικά αξιοκαταφρόνητα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το είδο τις μεταφορές. Ακολούθησα πολλές από τις προτάσεις των συναδέλφων και στι συμβαστικέ λύσει που προτάθηκαν δεν κρατήσαμε την μνήμα στο 20% της συνολικής απόστασης ούτε στην ε, γραμμή της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις διαδρομές την απόσταση των οδικών μεταφορών. Αυτές είναι δύο διαγραφές από τον οποίον ε, συμφωνήσαμε και νομίζω ότι και από αυτήν την αλλαγή καταλαβαίνουμε ότι και από τη δική μου την πλευρά υπάρχει διάθεση να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να είναι αντικείμενο συνένεσης και να το στηρίζουν όσο τα δυνατόν περισσότεροι. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό το στοιχείο του ορισμού. Το συζητήσαμε αρκετά αλλά παρόλο που πρέπει να καταλήξουμε, θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο περιθώριο για να μπορούμε πότε να, δίνουμε το χρόνο να φτάνει κανείς στους σταθμούς. Μετά ένα άλλο λεπτό θέμα είναι αυτό του καμποτάζ και της ανάπαυσης, της απόσπασης των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει να δούμε πώ θέλουμε να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες και στου ενδιασμένου τρόπου μεταφορών Μπα στο άρθρο 4. Είναι σημαντικό το θέμα των κινήτρων. Κινητρά που θα πρέπει να δίνουν τα κράτη-μέλη και το τι διευκολύνσει θα υπάρχουν. Αύριο ελπίζω θα πετύχουμε ευρεία πλειοψηφία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τι σχετικέ διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και να αποστείλουμε και ένα θερτικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τον κλάδο αυτό. Είναι σημαντικό για τη διατροπικότητα των μεταφορών. Και επ' αυτών θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των υπόλοιπων σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστούμε κυρία Γιούτο. Κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, οι διατροπικές μεταφορές ε, είναι πολύ καλές εάν πραγματικά λειτουργούν καλά και αν δεν παραμείνουν ένα προϊόν εδώ αν θέλετε πολύ περιορισμένο. Οπότε σε κάθε περίπτωση και με αυτήν την θα μπορούσαμε και με αυτή την πρόταση θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο να καταστούν αυτέ οι διατροπικέ μεταφορέ πιο ελκυστικέ. Ε, έχουμε καταρχήν απλουστεύσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την πρόταση τη Επιτροπή, ενώ από την άλλη πλευρά ασκούμε πιέσει στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε πραγματικά χρήσιμα δεδομένα. Μετά από την έγκριση, τη θέσπιση αυτή τη οδηγία δεν μπορούμε να αναμένουμε βέβαια ότι όλα θα βελτιωθούν αυτόματα. Ε, δηλαδή οι επιδόσει του σιδηροδρόμου δρόμου των σιδηρομικρόλογων μεταφορών παραμένουν πολύ χαμηλότερε από ό,τι των οδικών μεταφορών. Και παράδειγμα, η οι υποχρεώσει, ε, για παράδειγμα των οδηγών των αμαξιστοιχειών ε, να ε, μπορούν να ομιλούν τη γλώσσα τη κάθε χώρα που περνούν και ούτω καθεξή είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνεχιστούν με αυτόν τον τρόπο. Εάν θέλουμε λοιπόν να περάσουν οι μεταφορέ από τι οδικέ περισσότερο προ τι σιδηροδρομικέ, τότε θα πρέπει να εργαστούμε επίμονα επί τη δημιουργία ενό ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου. Αυτή η οδηγία αποτελεί ένα χρήσιμο πρωτοβήμα, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω πολύ σύντομα ε, ότι στην Αμερική οι οδικέ μεταφορέ λαμβάνουν ενισχύσει προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν, αν θέλετε, να παραμένουν ανταγωνιστικέ σε σύγκριση με τι διατροπικέ μεταφορέ ενώ το αντίθετο συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη. Όμω θα ήθελα να τονίσω κάτι ακόμα, ότι η συνεργασία σε σχέση με του τελευταίου φακέλου για αυτό το ζήτημα έχει λειτουργήσει πολύ καλά διακομματικά, οπότε ε, πραγματικά ε, συγχαίρω για τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει και θα ήθελα να ε, υποστηρίξω το, την συνεχιζόμενη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τον συμβασμό τον οποίο επιτύχαμε. Ευχαριστώ. Όλους σοσιαλιστές. Ε, ε, αντικαθιστώ την συνάδελφό μου την κυρία Ισαμπέλα Ντεμόντελ, η κυρία Γκρασφάντερ Βαντερχάντς. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, συγκέντρια την κυρία Γιούτο και όλου του εισηγητέ που προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιου συμβιβασμού σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώ δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα ε, για να συζητήσουμε αυτό το πρώτο τμήμα του ε, πακέτου κινητικότητα. Ε, είμαι πεπισμένο ότι οι κανόνε εδώ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστεροι εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε την αυξημένη χρήση των διατροπικών μεταφορών. Σίγουρα μπορούν να επιτύχουν περισσότερε βελτιώσει σε ό,τι αφορά την αποσυμφόρηση των οδικών μεταφορών αλλά και τη μείωση των εκπομπών του δεξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πω η μείωση του ποσοστού και των συγκεκριμένων καλύψεων είναι ένα βήμα που στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ, θεωρώ πως ε, εδώ γίνεται ένα σωστό βήμα και νομοθετικά σε ό,τι αφορά και ε, τη μετάβαση προς τα ημιρμουλκούμενα 44 ετών. Επίσης, αν θέλουμε αυτές οι διατροπικές ε, μεταφορές να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να προβούν και εκείνα σε επενδύσεις. Γι' αυτό, λοιπόν, προτείνω ε, και στις δικές μου τροπολογίες σε μια εξαίρεση από τους κανόνες σε ό,τι αφορά στις ε, κρατικές ενισχύσεις ε, κατά 35% της συνόλου χρηματοδότησης του project. Και επιτρέψτε μου να κάνω τώρα και εγώ κάποια προσωπικά σχόλια. Όπως γνωρίζουμε, το ζήτημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αφορά κυρίως τις οδικές μεταφορές. Οπότε αυτή η πρόταση θα πρέπει να μας απασχολήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε και σε σχέση με αυτό να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά. Επίσης θα πρέπει να, οπωσδήποτε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, συμφωνώ και εγώ με αυτό, και η διαγραφή αυτού του της, ε, της αύξησης ε, κατά περισσότερα από 20% της, ε, του, του τμήματος οδικής μεταφοράς είναι κάτι το οποίο ε, χαιρετίζω. Βέβαια θα θέλαμε να είχαμε επιτύχει λίγο κάτι παραπάνω, αλλά πάντοτε εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με συμβιβασμό και αυτό είναι το συμβιβασμό εμεί μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπελμπάου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Γιούτο για το έργο της όλο αυτό και την προσπάθεια φυσικά για την ε, συζήτηση και την ε, εκπόνηση των συμβιβασμών. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και με τις τροπολογίες μας που έχουν συμπεριληφθεί. Υποστηρίζουμε την απλούστευση, την ανάγκη εξορθολογισμού, καλύτερη πληροφόρηση, χρειάζεται και διαφάνεια, επίσης ενημέρωση και κάτι άλλο. Ε, να υπάρχει μια απέτηση συνοχής και συνέπειας. Μιλούμε για τις συνδυασμένες μεταφορές, λεγόμενες διατροπικές, και ποτέ δεν πρόκειται αυτές να είναι αποτελεσματικές αν δεν έχουμε συνέπεια στην εκτέλεση των έργων μας που σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δεσμεύσει, αλλά δεν εκτελούνται. Αρκεί να σκεφτούμε ε, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που δημοσιεύτηκε πριν από 15 μέρες, που τραβάει το αυτή σε όλα τα κράτη-μέλη, ακριβώς γιατί λείπει η συνοχή στην εκτέλεση των προγραμμάτων και των έργων αν θέλουμε να φύγουμε τα φορτηγά από τους αυτοκινητοδρόμους και πρέπει να φτιάξουμε σιδηρόδρομο μεταξύ άλλων. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις συνδυασμένε μεταφορές θα πρέπει να εκτελέσουμε τα έργα που εκκρεμούν. Και αυτό τονίζεται στην έκθεση για του συμβιβασμού. Είναι έξι στον αριθμό. Η ομάδα μας συμφωνεί με τους τέσσερις πρώτους. Αλλά είχαμε επιφυλάξεις ε, στη συνεδρίαση των σκιωδών για τις υπόλοιπε. η πέντε ε, συμβαστική πρόταση τη βάζει μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές σε τρία θέματα μόνο. Για μας αυτό είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει να είναι όχι υποχρεωτικό, αλλά να διευκολύνονται τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα και κυρίως τα κράτη-μέλη να δίνουν ε, κίνητρα με άλλες προτάσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται. Δεν μας φαίνεται σωστή αυτή η συμβαστική πρόταση έτσι όπως έχει συνταχθεί. Στη διάθεσή σας πάντως και μπορεί μέχρι αύριο να υπάρξει και κάποια αλλαγή. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Και για το συμβασμό 6 επίσης δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε μάλλον με τις κρατικές ενισχύσεις μέχρι ένα 35% τουλάχιστον δική μας ομάδα των φιλελευθέρων διαφωνεί. Από τους έξι βιβασμούς συμφωνούμε με τους τέσσερις μόνο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Monsieur Ευχαριστώ, κύριος Λούντγκρεν. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω αν σας διακόπτω. Τι έγινε. Αλλάξατε ομάδα. Έχετε το λόγο. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ ε, με πολλά από τα όσα ακούσαμε από την κυρία Γιούτο. Νομίζω πως ε, από ε, σε σχέση με τις περισσότερες πτυχές αποτελεί ένα καλό συμβιβασμό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλή δουλειά που κάνατε. Και νομίζω πως αυτά θα περιοριστώ. Δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί πραγματικά σε γενικές γραμμές θεωρώ πως είναι αρκετά καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Lundgren. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουντγκριν. Κύριε Νταλούντε, έχετε το λόγο. Tack för ordförande och tack till rapportören för ett gott eh, samarbete. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Εμείς θα θέλαμε η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εστιάσει περισσότερο στη σύγκληση προς την οικολογία. Υπάρχουν πολλά θέματα που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να φύγουμε από τον αυτοκινητόδρομο και να πάμε στις εσωτερικές πλωτές οδούς, ε, ε, στο σιδηρόδρομο και στις συνδυασμένες μεταφορές. Ε, στις συμβαστικές προτάσεις αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς να μιλάμε για τερματικούς σταθμούς ε, μεταφόρτωσης, αλλά και για πλατφόρμες διατροπικών μεταφορών και συνδυασμένων. Θα πρέπει να τα λέμε πολύ ξεκάθαρα και για το καμποτάζ και για τις διάφορες άλλες μορφές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ντέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην εισηγήτρια και την νομική υπηρεσία και έχει να κάνει αυτό με το συμβιβασμό Υπεριθμών διότι αυτή η συμβαστική πρόταση προεξοφλεί ε, το περιεχόμενο του λέξε Specialis και το θέμα για το καμποτάζ που την περασμένη εβδομάδα δυστυχώς ναυάγησαν στην Ολομέλεια. Και το περιεχόμενο ε, της ε, συμβαστικής πρότασης 4 συνάδει με τα όσα προτείνει η Επιτροπή Μεταφορών για το Lex Specialis και το Καμποτάζ, αλλά ξέρουμε ότι ακριβώς αυτή η θέση ιτήθηκε ε, και κατέπεσε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα λοιπόν είναι λάθος αυτή η αναφορά. Και από τη νομική σκοπιά επίσης δεν μπορώ να δεχθώ ότι έχουμε κάτι στο συγκεκριμένο φάκελο που κανονικά δεν έχει τη θέση του εδώ. Θα πρέπει αλλού να ρυθμίζεται αυτό και να αναφέρεται. Άρα, η συγκήτρια Ισκιώδης μαζί με το Συμβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τελειώσουν το τριμερή διάλογο και να συμφωνήσουν για αυτό το θέμα. Αλλά θα μας καθυστερήσει αυτό που έχει να κάνει με το Lex Specialis και το Καμποτάζ. Ρωτώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί αύριο θα ψηφίσουμε, αλλά έχω μεγάλα νομικά προβλήματα, αν το δούμε έτσι από την τυπική σκοπιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Εάν μου επιτρέπετε να απαντήσω στον κύριο Ντελή, δεν υπάρχει πρόβλημα Συμβατότητα. Διότι θα υπάρξει και πολιτική και νομική συμβατότητα η αβεβαιότητα είναι τελείως σχετική. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση που πάει στην ίδια κατεύθυνση με τις παρατηρήσεις του, της σκιώδους συγγετριάς μου, της κυρίας Ισασκούν. Η ομάδα FTD που συνήθως είναι καχύποπτη προς την Ευρώπη, για να το πω έτσι, σε σχέση με την δική μου την ομάδα που είναι τελείως ευρωομοσπονδιακής διάθεσης ίσως να μας πει τι θέση έχει σε σχέση με τις εθνικές μας ρυθμίσεις ε, ε, για τις μεταφορές. Εδώ μου φαίνεται πολύ αντιεπικουρικά όλα αυτά που προτείνονται. Θα πρέπει λοιπόν να μένουμε και σε ένα τοπίο πραγματικότητας, διότι ως ειδική της επικουρικότητας ήθελα να κάνω και αυτή την παρατήρηση σε σχέση με τις συμβαστικές που ανέφερε η κυρία Μπιλμπάου. Είναι ιδιαίτερα παρεμβατική ως προς τους εθνικούς κανόνες. Εδώ φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια αντιστροφή των πολιτικών ε, τοποθετήσεων που φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Κυρία Κουσέντσκα. Τώρα το λέω ωραία το όνομά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσουμε για την έκθεση και τις συμβαστικές τροπολογίες για τις μεταφορές τις συνδυασμένες, τις διατροπικές. Να πω ότι η συγκεκριτή έχει κάνει διεξοδική δουλειά στο θέμα. Και από όλους τους υπόλοιπους ακούω μια πολύ σαφή κατανόηση για τη συνολική πολιτική προτεραιότητα που υποκινεί την πρόταση αυτή, δηλαδή να κινηθούμε σε περισσότερη προσπάθεια οι εμπορικές μεταφορές να γίνονται αντί, για τις, ε, μέσω των αυτοκινητοδρόμων με άλλες οδούς. Δεν είναι κάτι εύκολο να το πετύχουμε, διότι θα το είχαμε πετύχει ήδη εδώ και καιρό, αν ήταν τόσο εύκολο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια για μερικέ από τι συμβαστικέ τροπολογίε που έχει προτείνει η συγγήτρια σε συνεργασία με τι άλλε πολιτικέ ομάδε ως προς την, ε, περιορισμό της οδικής απόστασης. Καλωσορίζουμε τη συμβαστική που διευκολύνει την πρόσβαση στο κοντινότερο τερματικό σταθμό. Αυτό δείχνει και την ευρύτερη ευρωπαϊκή διάθεση για, τις, για τα τερματικά, για τους σταθμούς βεβαίως δεν θα πρέπει να περιορίσουμε ιδιαίτερα αυτή την οδική απόσταση, γιατί ακριβώς αν ε, ε, γίνει πολύ σύντομη η απόσταση, δεν θα αφήσουμε περιθώριο να πτυχθούν και τα λέει μεταφορών πέραν των οδικών. Εξού και η πρότασή μα. Και ακούγοντα τι εξηγήσει και τη στήριξη για τη διαγραφή για το 20% της συνολικής, του συνολικού περιορισμού της αποστάσεως που αναφέρατε πολλοί από εσά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέξουμε στην τελική εκδοχή της πρότασης να παραμείνει αναφορά στο κοντινότερο κατάλληλο σταθμό τερματικό, διότι αν τα χάσουμε όλα δεν θα έχουμε και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε σε σχέση με την τωρινή πραγματικότητα και τελικά όντως θα επιστρέψουμε και πάλι στις οδικές μεταφορές. Όλοι συμφωνούμε ότι αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε τις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει απλούστευση τα ψηφιοποίηση, σαφήνεια και ε, ότι τα έγγραφα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ολεύληπτα. Γι' αυτό είναι σωστές οι τροπολογίες που ε, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι συνδυασμένε μεταφορές δεν δυσχεραίνονται. Λόγω, για παράδειγμα, διαφορετικών ε, εθνικών μορφοτύπων και εντύπων που θα κάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών του ελέγχου, ας πούμε, συμπατότητας δυσκολότερα από τη σήμερα. θεωρούμε σκόπιμη την πρόταση να υπάρχουν αυστηρότερε υποχρεώσει για την υποβολή εκθέσεων σε σχέση με του εθνικού στόχου και ελπίζουμε ότι όταν αυτό θα αρχίσει να ισχύει, τα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν αυτή την επιταγή και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέγει ε, εκθέσεις γεμάτες από περιεχόμενο που θα μπορεί με χαρά να υποβάλει σε αυτό το κοινοβούλιο ε, και να τι παρουσιάζει σχόλια για τη συμβαστική 6 και άλλες τροπολογίες που αφορούν τις κατοικές βοήθειες. Αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να εκφράσω αντίρρηση σε σχέση με τις συμβαστικές λύσεις που προτείνει η συγγήτρια πρέπει να υπάρχει και νομική βάση για να γίνει αυτό. Διότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει κανονισμού με συνολικέ εξαιρέσει, ομαδικέ εξαιρέσει, αυτό να γίνεται μέσω τροπολογιών σε αυτή την οδηγία νομικώ δεν στέκεται. Δεν ευσταθεί. Γι' αυτή λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή σα να την απορρίψει. Και ίσω ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί και αυτό προέκυψε και δεν θα σα εκπλήσει η σχέση του φακελού με τον κανονισμό για τι οδικέ μεταφορέ. Για μα είναι σημαντικό να υπάρχει νομοθετική αντιστοιχία μεταξύ των ε, συνδυασμένων διεθνών μεταφορών και των ε, οδικών διεθνών μεταφορών. Διότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε δίκαιο ανταγωνισμό, θεμετό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αυτών τρόπων μεταφορά εμπορευμάτων. Γι' αυτό η τροπολογία 4 που αποσαφηνίζει ακριβώ αυτή την αντιστοιχία και επαναλαμβάνει ότι ο κανονισμός για τις οδικές μεταφορές ισχύει όπως ίσχυε πάντα, το είπαμε νομίζω επανειλημμένο. Η οδηγία για του συνδυασμένου τρόπου μεταφορών δεν αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για τι οδικέ μεταφορέ. Απλώ επαναλαμβάνει, ενισχύει και επανεπιβεβαιώνει την ε, ισχύ του ρυθμιστικού πλαίσιου για τι οδικέ μεταφορέ όπω έχει διαμορφωθεί. Ξέρουμε ότι συχνά συζητιέται και κάποιε φορέ παρανοείται ο στόχος αυτής της πρότασης. Η πρόταση όμως ακριβώς στοχεύει, παρόλο που δεν είναι και καταφρόνητος ο στόχος, να προωθήσει την, τις συνδυασμένες μεταφορές για τα εμπορεύματα. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τοποθέτησή της. Κυρία Γιούτο, έχετε πλέον την τελευταία λέξη. Παρακαλώ πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους και οδείς για τις παρεμβάσεις τους. Σε ό,τι αφορά το θέμα το νομοθετικό, ε, αποσαφηνίστηκε νομίζω, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να, είναι, να μην είναι πλήρες. Πάντοτε ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα για την απόσπαση για το καποτάζ, θα πρέπει να ισχύσουν όσα ούτως ή άλλως προβλέπονται. Εάν υπάρχει, όταν θα υπάρξει και η έγκριση της οδηγίας αυτής, το κείμενο όπως έχει διατυπωθεί δεν θα εμποδίσει στην ε, εφαρμογή των υπόλοιπων κανόνων. Σε ό,τι φορά τώρα το θέμα και τους ενδιασμούς περί αναλογικότητας και αν έχουμε καλύψει κάποια πράγματα ή όχι, μη σας εκπλήσει κύριε Ρικέ διότι στο κείμενο αφήνε, ε, αφήνεται μεγάλο περιθώριο δικαιωτική ευκαιρία στα κρατη να επιλέξουν ποιον τρόπο θέλουν να προωθήσουν. Θα πρέπει μάλιστα να δώσουμε κίνητρα στα κρατη Υπάρχει λοιπόν μία ε, βασική υποχρέωση να επιλέξουν κάτι. Δεν μπορεί ένα κράτο μέλο να μην ε, Μάλλον, αν ένα κάτω μέλο δεν έχει κίνητρο, δεν θα έχει και λόγο να πάει προ έναν τρόπο μεταφορά. Έχουμε λοιπόν ελευθερία επιλογή για τα κράτη. Αλλά τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να επιλέξουν κάτι. Οφείλουν να επιλέξουν, αλλά μπορούν να επιλέξουν από ένα μεγάλο φάσμα επιλογών. Αυτή είναι η δική μα προοπτική. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιούτο. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 9. Και να συνεχίσουμε με την έκθεση του κυρίου Ντελή. Προώθηση των ε, καθαρών και ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ντελή και θα δώσω το λόγο και στους συνεισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και βεβαίως θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος. Κύριε Ντελή. Merci, Madame la Présidente. Actually... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε εδώ μια νομοδότηση από την πλευρά τη ε, δική μα επιτροπή ε, που καταφέραμε τελικά να την κλείσουμε πριν από την ε, χθεσινή, ε, από την αυριανή συγγνώμη, προθεσμία. Και έχουμε λάβει 252 τροπολογίε συνολικά από του συναδέλφου. και τις περισσότερες από αυτές μπορέσαμε να τις συμπεριλάβουμε σε 21 συμβαστικές τροπολογίες. Ε, σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, από κοινού με τους κοιόδες συζητητές, ε, νομίζω πως ε, καταφέραμε να, να τηρήσουμε τους βασικούς στόχους ε, που είναι καταρχήν η τεχνική ουδετερότητα και η διεύρυνση δηλαδή τη οπτική γωνία τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτή την τεχνική ιδιαιτερότητα. Από εκεί και μετά, εκείνο που προσπαθήσαμε επίση να διαφυλάξουμε σε αυτέ τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε είναι ένα έδο ασφαλεία ε, δικαίου, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση αυτή τη οδηγία ε, με την οδηγία για την υποδομή των εναλλακτικών καυσίμων και τα είδη των καυσίμων. Και επίση προσπαθήσαμε εδώ να θέσουμε ρεαλιστικού στόχου σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη και κατά συνέπεια και τις ε, σχετικές υποχρεώσεις που θα βαρύνουν τους Δήμους και τις κοινότητες και τις άλλες ε, περιφερειακές αρχές ε, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει έτσι ώστε να επιτευχθούν τα ε, νούμερα τα σωρευτικά σε εθνικό επίπεδο. Και επίση ε, καταφέραμε εδώ να συμπεριλάβουμε και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πράγμα αποτελεί μια καινοτομία, καθώ η αρχική πρόταση τη Επιτροπή δεν τα συμπεριλάμβανε αλλά και εμεί έχουμε, για παράδειγμα, τι διάφορε υπηρεσίε οδήγηση, δηλαδή του σοφέρ και ούτω καθεξή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε έχει νόημα να συμπεριληφθούν και αυτέ οι υπηρεσίε εδώ ε, στο πεδίο εφαρμογή. Ε, και επίση έχουμε διευρύνει λίγο το πεδίο εφαρμογή, γιατί έχουμε περιλάβει νέε κατηγορίε οχημάτων, όπω την κατηγορία ε, λάμδα των μηχανών, των δικύκλων δηλαδή αλλά και κάποιες ακόμα ε, υπηρεσίες μεταφορών, για παράδειγμα όπως ε, ε, μεταφοράς δεμάτων ε, ή συλλογή απορριμμάτων εφόσον έχουν δημοσιο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν νομίζω πως το, αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές ε, που ήταν ανοιχτοί ε, σε όλες τις προτάσεις που έκανα και νομίζω πως πραγματικά φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και κατά συνέπεια ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλη. Αρχίζει η συζήτηση. Κυρία Άντερσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την ε, σκληρή δουλειά που έκανε εδώ και όλη η ομάδα του. Γιατί και εγώ συμφωνώ ότι πραγματικά έχουμε καλό αποτέλεσμα το οποίο απηχείται και από ε, την ευρεία συνένεση που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στι διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Ε, σε ό,τι αφορά τι θετικέ πτυχέ αυτού του συμβασμού, ε, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ότι δηλαδή είναι πολύ καλό καταρχήν το γεγονό ότι έχουμε διευρύνει το πεδίο εφαρμογή ε, και επίση είναι πολύ χρήσιμη και η τροπολογία σε ό,τι αφορά ε, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ειδικέ υπηρεσίε εκεί. Χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο. Ε, από μια άποψη θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί λίγο πιο μακριά ακόμα, γιατί εδώ έχουμε και σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, τα κινητά μηχανήματα, δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται στο κατασκευαστικό τομέα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πρόκειται για ένα δύσκολο τομέα από τεχνική άποψη, οπότε όπως η Επιτροπή θα συνεχίζει να εξετάζει αυτό το ζήτημα στο μέλλον. Επίση, ε, θεωρώ πω ε, είναι καλέ οι βασικέ τροπολογίε που επιτύχαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και μία ρήτρα αναθεώρηση σε αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε αλλά και προκειμένου να υπάρχει μια εκτελεστική πράξη η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να προβαίνει σε ενημερώσεις ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ε, εγώ δεν ήθελα να, είμαστε, να επιμείνουμε τόσο πολύ στον ορισμό των εναλλακτικών καυσίμων, γιατί ορισμένα από αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πραγματικά χρησιμεύουν για τα καθαρά εντό εισαγωγικών οδικά οχήματα, αλλά προ το παρόν μπορώ να το αποδεχτώ. Ελπίζω πω η δουλειά μα θα συμβάλλει στη συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή ΕΝΒΗ ε, και γνωρίζω πω θα γίνει ένα ενδιαφέρον διάλογο εκεί. Ε, επιχαίρω το γεγονό ε, ότι Εμεί ακολουθήσαμε μια τόσο επικοδομητική και θετική προσέγγιση από πλευρά της Επιτροπή Τρένα. Ευχαριστώ. Κύριε Λούντκρεν, θέλετε να πάρει το λόγο, όχι. Κύριε Νταλούντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους όσοι ε, συνεισέφεραν στην προσπάθεια αυτή, εξαιρετική συνεργασία. Εμείς επιθυμούσαμε όμως η Επιτροπή μας να είναι πιο φιλόδοξη οδηγία αυτή θα πρέπει να μας βοηθήσει για να έχουμε περισσότερη εφορία και βιωσιμότητα στον κλάδο των μεταφορών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εμείς δεν ακολουθούμε ε, την αγορά. Ε, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Την επόμενη δεκαετία θα είναι τεράστιες ε, ε καινοτομίε και οι εξελίξεις και η καθαρή κινητικότητα είναι πραγματικά μια πρόκληση για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά το, το λεγόμενο retrofitting που είναι η ανακαίνιση και η ε, βελτίωση, ε, κανονικά θα πρέπει να αποσύρονται και να διαλύονται και να καταστρέφονται τα οχήματα αυτά παρά να προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο και Επίσης, ε, οι καταληκτικές προθεσμίες ε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ε, για να σταματήσει να καταργηθεί το retrofitting. Και, μας ενδιαφέρει καθαρή κινητικότητα και όχι αυτές οι εμβαλωματικές λύσεις. Για την κατηγορία L, τα τετράτροχα οχήματα, θα πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρή ρύθμιση και ε, η νομοθεσία να εφαρμόζεται και να ε, μεταφέρεται ταχύτερα σε εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ κύριε Νταλούντε. Κυρία Κίλονεν, ναι, ναι, θέλετε να πάρετε το λόγο. Alors, me Ωραία. Ε, στρέφομαι μέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπέλ Βαντόρν. Παρακαλώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαιρόμαστε για την ευρεία αποδοχή που γνώρισε και υποστήριξε η πρότασή μας. Φαίνεται ότι όλοι θέλουν να διαβεβαιωθεί το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, ε, Θα πρέπει να δώσουμε ένα κοινό κανονισμό, ε, ορισμό μάλλον του καθαρού οχήματος και οπωσδήποτε να έχουμε στόχους ε, κατώτατου. και σε σχέση με τα όσα είπαν οι τελευταίοι ομιλητέ, ε, πρέπει να δείξουμε και μεγαλύτερη φιλοδοξία. Τι κρατάμε από τις διάφορες συζητήσεις, γιατί έχουμε σύγκρατηση, ότι χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα ως προς τον ορισμό, το, το επίπεδο των στόχων και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν αυτοί. Για τον ορισμό του καθαρού οχήματο, αυτός θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να βασίζεται ε, στα οριακές τιμές για την εκπομπή καυσαερίων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα βαρέα ε, επαγγελματικά οχήματα, Όπως είδατε, ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να, παίρνουμε, να πάρουμε την απόφαση γιατί δεν έχουμε τις τεχνικές εκείνες τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε. Θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι πηγαίνουμε γενικώ προς σωστή κατεύθυνση με βάση την πρόταση που βρίσκεται επιτάπητος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντέλη, έχετε το λόγο για να κλείσετε. Thank you, uh, uh θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια που κάνατε. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ακόμα πιο φιλόδοξοι, ή τέλος πάντων όσο πιο φιλόδοξη γίνεται, αλλά ο στόχος θα πρέπει να είναι να συμμετάσχουν εδώ ε, οι ε, κυβερνήσεις και οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και το νωρίτερο δυνατό. Γιατί μπορούμε να έχουμε ό,τι πιο φιλόδοξο μπορούμε επί χάρτου, αλλά αν τελικά δεν αναλάβουν τη δέσμευση από την πλευρά του τα κράτη-μέλη και διάφορες τοπικές αρχές, δεν θα επιτύχουμε κάτι και γι' αυτό ε, χαίρομαι για το ότι όλοι κατάφεραν να αποδεχτούν αυτή την προσέγγιση και κατά συνέπεια ε, προσπάθησαν ε, μαζί μου να βρούμε μια ρεαλιστική αφενός αλλά και φιλόδοξη προσέγγιση αφετέρου. Οπότε σας ευχαριστώ όλους και θα σας δω και πάλι αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλη. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο σε 9 ώρα το πρωί. Λήξεις λοιπόν του πρώτου τμήματος της ε, σημερινής συνεδρίασης και θα παρακαλέσω όλους ε, όσοι δεν είναι συντονιστές και δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται. Και συντονιστές ελάτε στις 5.30, ένα τέταρτο νωρίτερα. 5.30 ώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Υπόλοιποι αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ.